Uh, um, Καλημέρα σε όλους. Όπως βλέπετε, είμαι πανευτυχής που ο ε, Πίτροπος Μίμητ είναι ήδη εδώ. και προσελκύει πολύ τις κάμερες των φωτογραφικών μηχανών. Ελπίζω να βγω κι εγώ σε καμιά γωνίτσα, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ τους εκπρόσωπους του τύπου να καθίσουν να, και για να βλέπω και του υπόλοιπου ευρωβουλευτές. Και εκείνοι θέλουν να τους βγάλετε καμιά φωτογραφία ο, πριν φύγετε. Λοιπόν, ωραία, όλα έχετε βάλει τα καλά σας. Πολύ ωραία, ας ξεκινήσουμε. Δεν βλέπω κυρίες φωτογράφους εκεί πέρα πίσω. Όχι, ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση που είναι η Επιτροπή Ακρόασης του οριστέντος επιτρόπου της Κροατίας για την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η μέρα σήμερα για το Κοινοβούλιο και για την Ευρώπη και είναι μεγάλη μου τιμή που προεδρεύω σήμερα είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε χρήσιμη και επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τον Οριστέντα Επίτροπο. Επίσης ε, θα ήθελα να καλωσορίσω επισήμως τους Κροάτες Διερμηνείς, γιατί και πάλι είναι η πρώτη επίσημη ευκαιρία όπου θα έχουμε Κροάτικα στην συνεδρίαση. Είστε πάνω εκεί κάπου, εσείς θα τους χαιρετήσετε βέβαια και θα τους πει, εγώ δεν τους βλέπω γιατί είναι λίγο πίσω μου. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς θα τους χαιρετήσετε και θα τους πείτε πόσο ευπρόσδεκτοι είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν ξεκινήσουμε την ε, συνεδρία, θα ήθελα να κάνω κάποιες επίσημες ε, παρατηρήσεις για την διοργάνωση της ακρόασης, για τις ευθύνες του αρμοδιότητες του Επιτρόπου και κάπως το ιστορικό πριν ξεκινήσουμε. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω το ακροατήριό μας στο διαδίκτυο όπου αναμεταδίδεται ζωντανά η συνεδρίαση αυτή, όπως και όλες οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Να καλωσορίσω όλους όσους παρακολουθούν στο διαδίκτυο και ίσως και νέους κροατές ή θεατές ε, στην Κροατία. Και δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να πω άλλη μια φορά πως όλες μας οι συνεδριάσεις ε, αναμεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο και είστε ευπρόσδεκτοι να τις παρακολουθείτε. Ε, ελπίζω πως θα εκτιμήσετε τη δουλειά που κάνουμε για τους καταναλωτές και υπάρχει και ένα δελτίο τύπου που ενημερώνει για τη δουλειά μας. Μπορείτε να, το, να γίνετε συνδρομητές και να λαμβάνετε τα mail. Ε, μετά από αυτά, ε, αυτή την ε, πρώτη παρουσίαση να προχωρήσουμε στις εργασίες μας. Σε αυτή η συνεδρίαση γίνεται από κοινού με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, διότι μάλλον και ο πρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, μου το ζήτησε και έτσι τρεις ευρωβουλευτές, η κυρία Κλάς, θα είναι εδώ ω αναπληρώτρια αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο με άλλε τρει ευρωβουλευτέ, ώστε να θέσουν ερωτήσει σε σχέση με τι αρμοδιότητε του Επιτρόπου που αγγίζουν και τα θέματα υγεία, ιδιαίτερα το θέμα που αφορά το ιατροτεχνικό, ιατροτεχνικά προϊόντα γιατί μέσα στο χαρτοφυλάκιο των αρμοδιοτήτων του κυρίου Μίτσα, αν τελικά εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, όλα αυτά θα σχετίζονται, θα με την ε, ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτή, θέματα για τα οποία εμείς εργαζόμαστε, καθώς και θα έχει σημαντικές ευθύνες για, τα, για προϊόντα υγείας. Και φυσικά αυτή είναι η βασική εργασία της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και προστασία του καταναλωτή. Σύμφωνα τώρα με την, ε, τον εσωτερικό μα κανονισμό, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει του οριστέντε επιτρόπου επί τη βάση των γενικών του ε, προσόντων, τη ευρωπαϊκή του προσήλωση ε, και τη προσωπικότητά του, αλλά και τις γνώσεις του για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, καθώ και τι επικοινωνικέ του ικανότητε. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό είναι αυτό που έχετε υπόψη σα και εσείς και ο Επίτροπος καλείται να υποβάλει ένα προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο που όλοι έχετε στους φακέλους σας και ξέρω πως ήδη θα το έχετε μελετήσει και οι γραπτές απαντήσεις ε, σας έχουν δοθεί σε όλες τις γλώσσες. Επίσης έχετε τη δήλωση του Επιτρόπου προσωπικών ε, διαφερόντων και συμφερόντων και βλέπω εδώ και τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που υπ' αυτή τη διαδικασία έχει την αρμοδιότητα να, εκφρα... να εξετάσει τον κώδικα διοντολογίας, να τον ελέγξει και να κάνει παρατηρήσεις αν έχει. Και αυτή είναι επίσημο... επισήμως υποχρέωσή μας. Τώρα όσον αφορά την ακρόαση, το χρονοδιάγραμμά μας θα είναι πολύ αυστηρό το πρόγραμμά μας σήμερα. Θα δείτε λοιπόν διαρκώς το χρονόμετρο να, να δουλεύει, γιατί θέλουμε όσο γίνεται περισσότεροι οι ευρωβουλευτές να θέσουν ερωτήσεις και να ε, κρατήσουμε την ώρα δίκαια. Γι' αυτό θα λειτουργήσουμε ως εξής. Ε, συντόμως ε, θα καλέσω τον Οριστέντα Επίτροπο να προβεί σε μια εναρκτήρια δήλωση, όχι πάνω από 10 λεπτά. Το υπόλοιπο του χρόνου μας, 2,5 ώρες, θα είναι ερωταπαντήσεις. Θα ξεκινήσουμε με όλες τις πολιτικές ομάδες και τους συντονιστές τους που θα υποβάλλουν ερωτήσεις ο έκαστος και έπειτα θα έχουν και ευκαιρία για συμπληρωματική ερώτηση, για επερώτηση. Και να θυμίσω στους συναδέλφους και στον Επίτροπο πώς θα δουλέψουμε. Έχετε maximum ένα λεπτό για μια πρώτη ερώτηση. Ελπίζω, Γιάννη, πως θα έχετε μία ερώτηση ψηλής ποιότητας. Ορισμένοι συχνά έχουν δύο ερωτήσεις και λαθ λαθρέω, ε, εισάγουν και μια τρίτη. Ε, ο υποψήφιος επίτροπος θα έχει δύο λεπτά για να απαντήσει και αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε το, το πλεονέκτημα της επερότασης έχετε 45 δευτερόλεπτα. Να σας θυμίσω όμως και είμαι πολύ αυστηρός από αυτό όπως θα θυμάστε και από παλιότερες ακροάσεις οι επερωτήσεις θα πρέπει να σχετίζονται με το θέμα της αρχικής σας ερώτησης. Και αν προσπαθήσετε λαθρέα να κάνετε μια ακόμα ερώτηση θα σας κόβω το λόγο γιατί δεν είναι δίκαιο για τους υπολείπους. Και έπειτα ο υποψήφιο επίτροπος έχει ένα λεπτό για την επόμενη ε, απάντηση. Λυπούμε που είναι όλα έτσι πολύ τυπικά, αλλά μόλις θα πάρουμε το ρυθμό μας θα δείτε ότι λειτουργούν όλα πολύ καλά. Να σα θυμίσω στους συναδέλφους επίσης ότι αναμένω οι ερωτήσεις προ τον επίτροπο να εστιάζονται στα θέματα για τα οποία θα είναι υπεύθυνο. Ξέρω πως είναι μέρος του ευρύ, της ευρύτερης ομάδας του συλλογικού οργάνου και θα, θα, θα εργάζεται επί διαφόρων οριζοντήρων θεμάτων. Να σας θυμίσω πως ο οριστής επιτροπός δεν έχει αναλάβει ευθύνη όσον αφορά τα τρόφιμα ή την ασφάλεια των τροφίμων, ούτε το καπνό, ούτε τα θέματα που αφορούν δημόσια υγεία. Αν μπορείτε με κάποιο κομψό τρόπο να βρείτε ώστε να το συνδέσετε με την επικαταναλωτική πολιτική, καλώς. Αλλά ερωτήσεις που δεν αποτελούν κομμάτι του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου δεν θα τις επιτρέψω. Και αυτό προσχάρει χάρη δικαιοσύνης απέναντι σε όλους. Εντάξει, τώρα κάνω τον τελετάρχη λίγο, με συγχωρείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω πως θα μπορέσουμε έτσι να αποκομίσουμε τα μέγιστα ωφέλη από αυτή την ακρόαση, να ελέγξουμε τις γνώσεις του Επιτρόπου επί του χαρτοφυλακίου του. Σας καλώ λοιπόν αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Νομίζω πως σας θύμισα όλα στις λεπτομέρειες. Έχω, έχουμε διερμηνία στις 23 γλώσσες τώρα, τις 22 που είχαμε συγκροατικά. Και νομίζω πως τα υπόλοιπα θα κυλήσουν ομαλά. Ας προχωρήσουμε. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν, καλώ τον οριστέντα επίτροπο να μας απευθύνει το λόγο για πρώτη φορά στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Με μεγάλη χαρά και τιμή εμφανίζομαι σήμερα ενώπιό σας και αναζητώ την έγκρισή σας για να είμαι το πρώτο μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Κροατία αισθάνομαι μεγάλο προνόμιο που έχω οριστεί ως Επίτροπος για ε, πολιτική προστασία των καταναλωτών. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να ε, γίνει διαφορά και με πολύ θετικό τρόπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Εάν οριστώ και επιβεβαιωθώ, θα επιζητήσω στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Έχουμε κοινά συμφέροντα, βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε καλύτερη ευκαιρία να το πράξουμε αυτό και πιθανότητες εάν συνεργαστούμε. Για το λόγο αυτό θα επιζητήσω το διακομματικό τρόπο συνεργασίας πέρα από πολιτικές ε, ομάδες και εθνικότητες. Επιτρέψτε μου τώρα να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Ως πρώτος οριστής επίτροπος έχω την ευκαιρία να μιλήσω κροατικά. Μπορεί να μην είναι ιστορία εν το γεννάστε, αλλά μπορεί να είναι ιστορία εν το ακροάστε. Χαιρετίζω λοιπόν την ευκαιρία που έχω να μιλήσω τη γλώσσα μου. Ε, Κροατία ε, βεβαίω ενδιαφέρεται για μεγάλη προστασία των καταναλωτών και χρειάζεται αλληλεγγύη όλων μεταξύ αυτών και του νέου Επιτρόπου, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα των δύο Επιτροπών που θα δώσουν μια νέα πνοή στην ε, οικονομική και κοινωνική συνεργασία και με τους καταναλωτές για την προαγωγή της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε κοινέ αξίες, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να τις διατρανώνουμε και να τις υπηρετούμε ιδιαίτερα στο παρόν οικονομικό πλαίσιο που θα πρέπει ε, να ανταποκριθεί η Ευρώπη σε μεγάλες οικονομικές προκλήσεις. Η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία διέπουν επίσης και την πολιτική προστασία καταναλωτών. Και αυτές οι αξίες με ενέπνευσαν όταν στην Κροατία προώθησα το πρώτο νομοθετικό πακέτο και τη δέσμη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών. Επίσης ενθαρρύνω και ενθάρρυνα τους ε, Κροάτες ε, καταναλωτές να υποφεληθούν από αυτές τις δυνατότητες. Ποια είναι τα βασικά σημεία. Μεγάλη πρώτη οικονομική διάσταση που απορρέει από την οικονομική ισχύ που έχουν οι καταναλωτές. 56% του ΕΕΠ είναι οι δαπάνες των καταναλωτών στην Ευρώπη, άρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, την αναζωογόνηση της οικονομίας και ε, στην καινοτομία και στην αηφορία. Οι καταναλωτές έχουν κεντρικό ρόλο για την ανάπτυξη του πραγματικού δυναμικού της ενιαίας αγοράς. Άλλωστε αυτό το λέει και η πράξη για την ενιαία αγορά. Αλλά οι καταναλωτές δεν είναι μόνο αγοραστές. Υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση στην πολιτική των καταναλωτών που είναι η κοινωνική διάσταση συγκεκριμένα ωφέλη και ευεργετήματα επιζητούν οι ίδιοι οι καταναλωτές και θα πρέπει οι αγορές να εργάζονται υπέρ των καταναλωτών και όχι το αντίστροφο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα αυτό που οι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται σε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. Θα πρέπει να ε, πιάνει ε, τόπο κάθε ευρώ, κάθε κούνε οποιοδήποτε άλλο εθνικό νόμισμα. Η πολιτική των καταναλωτών θα πρέπει να δίνει ε, την εξουσία στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερες αγορές, να εξοικονομούν τα χρήματά τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με τρόπο αποτελεσματικό. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, εγώ είμαι ρεαλιστής. Το υπόλοιπο της ιδέας της παρούσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μεν περιορισμένο, πλην όμως επαρκές για να έχουμε πραγματική ε, πολιτική με επιπτώσεις και να δείξουμε πρακτά, ε, πρακτικά συγγνώμη, αποτελέσματα. Ε, θα εργαστώ προς την ατζέντα του Ευρωπαίου Καταναλωτή που έχει διαμορφωθεί ουσιαστικά και από το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή σας. Ε, μ' αρέσει αυτή η συνολική προσέγγιση. Θα ε, εργαστώ ως θεματοφύλακα της ατζέντα αυτή σε συνεργασία με άλλους επιτρόπους, ιδιαίτερα την Αντιπρόεδρο Ρέντι, ε, υπό συνεχή παρακολούθηση. Ως βασική μου προτεραιότητα θα έχω τα εξής. Εδραίωση, συνεργασία, επικοινωνία. Πρώτον, για να ε, κατοχυρωθεί και να ιδρυωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχουν ε, εκρεμείς νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ιδιαίτερα για τις ε, ιατροτεχνικές συσκευές και ιατροδιαγνωστική, για την ασφάλεια των προϊόντων και τις τραπεζικές καταθέσεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να εγκριθούν αυτά τα τρία κατά τη διάρκεια της παρούσης θητείας. Και όπου είναι ήδη εγκεκριμένη νομοθεσία θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή και αποτελεσματική μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, την εκάστοτε και εφαρμογή ε, νέες διατάξεις επίσης ε, για τα καλλιντικά ε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Στη συνεργασία με τους ενεχομένους θα επενδύσω πάρα πολύ. Η προστασία των καταναλωτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες πολιτικές και άλλους τομείς πολιτικής και θα πρέπει να υποστηρίζεται ένεργα από διάφορους ε, φορείς και εταίρους. Ε, θα αφιερώσω πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό, αρχής γενομένης βεβαίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα εκπροσωπώ στο Κολέγιο των Επιτρόπων, στο Σώμα των Επιτρόπων του καταναλωτές και θα επιζητήσω ισχυρές συμμαχίες με άλλους ε, επιτρόπους που άπτονται τα χαρτοφυλάκια τους στα θέματα των καταναλωτών. Προσβλέπω και σε πρωτοβουλίες υπέρ των ε, καταναλωτών ε, διαμέσου άσκησης πολιτικής. Ως δημοκρατικά εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, εσείς οι βουλευτές για μένα θα είστε σημαντικοί εταίροι, ιδιαίτερα οι δύο επιτροπές που συνδιοργανώνουν τη σημερινή ακρόαση. Η ε, πολιτική των καταναλωτών είναι πολιτική των λαών και ο λαός είστε εσείς θεωρώ τις ε, ενώσεις καταναλωτών ως σημαντικό συνδετικό κρίκο με τους καταναλωτές. Βέβαια αυτό είναι κύρια ευθύνη των κρατών μελών ε, να λειτουργούν σωστά τέτοιες ενώσεις και οργανώσεις σε κρατικό επίπεδο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δώσει πολύτιμη βοήθεια και με χαρά να συνεισφέρω. Θα πρέπει επίσης να συνεργαζόμαστε με διεθνείς εταίρους όπως είναι η Κίνα. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτό για να βεβαιωθούμε ότι όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας και μάλιστα στην πηγή. Συνεργασία με τη βιομηχανία για ουσιαστική υποστήριξη των καταναλωτών και ανταγωνισμός να είναι επίσης όρης. Αυτά είναι οι διόψεις του ίδιου νομίσματος. Ε, έτσι λοιπόν θα συνεργαστώ με τη βιομηχανία με τρόπο διαφανή και ειλικρινή. Κυρίες και κύριοι, η συνεργασία έχει ιδιαίτερη σημασία για την εφαρμογή και την υλοποίηση και την επιβολή των νόμων. Εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα πριν τα τέλη του 2013. Ε, δικαιώματα καταναλωτών που δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά ακυρώνονται. Και ε, η επιβολή και η εφαρμογή γίνεται κυρίως σε εθνικό επίπεδο και στην αγορά. Αλλά μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις εθνικές προσπάθειες. Αυτό έχει γίνει ε, πολύ αποτελεσματικά μέσω του αντιστοίχου δικτύου ε, και ε, στόχος μου είναι να το προωθήσω έτσι περαιτέρω. Θέλω να δω πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δίκτυο για ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μπορούν να διευρυνθούν οι τομείς που καλύπτονται. Μπορούμε να ορίσουμε βέλτιστες πρακτικές, να τις ανοιχνεύσουμε. Θα πρέπει να δούμε πολύ σύντομα τα αποτελέσματα και πολύ ε, σύντομα επίσης ε, ήθελα να δω την αντίστοιχη έκθεση που ε, προετοιμάζεται και αναμένεται να κατατεθεί του χρόνου. Να δούμε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο και αν ε, δίνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ε, θέλω να προβληματιστούμε μαζί ε, με εσάς και άλλους εταίρους στους επόμενους μήνες για αυτά τα θέματα. Κυρίες και κύριοι, τρίτη μου προτεραιότητα είναι η ενεργή και ορατή προώθηση και προβολή και επικοινωνία για την πολιτική καταναλωτών στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να διαδώσουμε τι κάνουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό ε, χρειάζεται πιο στοχευμένη πληροφόρηση των καταναλωτών με σαφή γλώσσα και απλή για να καταλάβουν οι πολίτες και να έχουν στοιχεία, αλλά να έχουν και την εμπιστοσύνη ότι προστατεύονται και ότι έχουν δικαιώματα που μπορούν να τα επικαλεστούν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για καταναλωτέ που ζουν σε χώρες ε, με ασθενή μάλλον καταναλωτική ε, κουλτούρα. Και υπάρχουν τομείς που μπορούν οι καταναλωτέ και χρήματα να εξοικονομήσουν και ενέργεια ε, να πληρώνουν χαμηλότερα τιμολόγια, καλά προϊόντα σε καλύτερες τιμές και καλύτερη ποιότητα. Θα χρησιμοποιήσω την εντολή μου έτσι ώστε να δημιουργήσω ε, μεγάλη συνειδητοποίηση ε, του κοινού και ενδιαφέρον για θέματα καταναλωτών. Εάν επιτύχουμε αυτό θα βοηθήσει να αποδείξουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης για τους πολίτες και αντίστοιχα μπορούν να τους ενθαρρύνει να ψηφίσουν του χρόνου στις ευρωεκλογέ, να προσέλθουν στις ευρωεκλογέ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πραγματικότητα μεταβάλλεται. Οικονομική κρίση, ψηφιακή επανάσταση, παγκόσμια αγορά. Θα πρέπει αντίστοιχα να προσαρμόζεται και η προστασία των καταναλωτών. Αν μου δώσετε την ευκαιρία, είμαι διατεθειμένος να αξιοποιήσω όλο αυτό το δυναμικό. Είναι μια πολιτική των πολιτών ουσιαστικά, αγγίζει την καθημερινή ζωή, συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση με του πολίτε τη συχνά ε, απαντά και στη βασική ερώτηση των Ευρωπαίων πολιτών, που είναι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε υποψήφιε Επίτροπε, για μια πολύ ολοκληρωμένη εισαγωγική παρέμβαση θα θέλαμε πρώτα να ακούσουμε τις ερωτήσεις ε, των συντονιστών της Επιτροπής και θα ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα Σουσφάπ. Ένα λεπτό για την ε, αρχική του ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μίμητσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Ε, θα ήθελα να ε, θέσω την ερώτησή μου. Μία από τις ε, προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία θα ανήκετε, αν επιβεβαιώσουμε την υποψηφιά σας, είναι η βελτίωση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, το είπατε και αυτό, και η Επιτροπή έχει υιοθετήσει ομόφωνα μία έκθεση για την εσωτερική αγορά, όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει ο Επίτροπος να κάνει περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν. Αναφερθήκατε στα sweeps και ε, στις ε, γραπτές σας ε, παρατηρήσεις έχετε πει ότι πιστεύετε στην καλύτερη εφαρμογή χωρίς νέα νομοθεσία. Αυτό μου φαίνεται πολύ λογικό, διότι πράγματι μερικές φορές το λιγότερο μπορεί να είναι περισσότερο, αλλά για τους λίγους μόνες μήνες της θητείας σας μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνετε συγκεκριμένα για να βελτιώσετε την εφαρμογή της νομοθεσίας για την αστερική αγορά, να είναι αυτό προς όφελος ε, των καταναλωτών. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα παραδείγματα που μπορείτε να ε, επεκτείνετε τα SWIPS ε, και που μπορείτε να φροντίσετε την εφαρμογή συγκεκριμένων νόμων. Ο υποψήφιος Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σβάμπ για την ερώτηση αυτή που μου επιτρέπει να αναπτύξω λίγο περισσότερο την γενική διαδικασία ε, διαμόρφωσης της πολιτικής που θεωρώ ότι είναι ε, καθήκον κλειδί του νέου Επιτρόπου. Ε, προσπάθησα να εξηγήσω ότι η πολιτική των καταναλωτών δεν είναι μια μεμονωμένη πολιτική, είναι οριζόντια, εγκάρσια και απαιτεί συνεργασία με όλους τους άλλους επιτρόπου, επιτρόπους στα θέματα όπου οι δικές τους δράσει μπορούν να επηρεάσουν τα συμφέροντα ή να καθορίσουν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Οι ενέργειές μου λοιπόν θα βασιστούν ε, στο θεματολόγιο που αφορά τους καταναλωτές θεωρώ ότι είμαι θεματοφύλακα ε, ε, των θεμάτων αυτών, του θεματολογίου αυτού, και το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να επικεντρωθώ στου τέσσερι πυλώνε. Ε, καταρχήν, ασφάλεια των προϊόντων. Αυτό είναι το κυριότερο και αυτό συνδέεται με τις με, τα προσόντα και δεξιότητες του νέου ε, Επιτρόπου. Προσλέπω στην καλή συνεργασία με την Επιτροπή σας και με τις δύο Επιτροπές σας για να ε, δούμε νομικές προτάσεις για, τα, για τις ιατρικές συσκευές, τα ιατρικά βοηθήματα, ε, το πακέτο ασφάλειας των προϊόντων ε, καθώς και την εποπτεία της αγοράς, καθώς ε, και τους ε, τραπεζικούς λογαριασμούς. Ελπίζω αυτά τα νομοθετήματα να εγκριθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας του Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν θα είναι μια πρώτη, νομοθετική, μια πρώτη σειρά νομοθετικών προτάσεων. Εάν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, θα επικεντρωθώ στην Ε, αναθεώρηση της ε, συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών. Θα ε, ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτά στα κράτη-μέλη και εάν δείξουν οι αναλύσεις ότι απαιτείται κάτι τέτοιο, θα καθορίσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο συντονισμού ε, για την εφαρμογή των ε, κανόνων που αφορούν τα προϊόντα. Επίσης μας ενδιαφέρει η ενδυνάμωση του καταναλωτή, η καλύτερη πληροφόρηση του καταναλωτή. Αυτό προφανώς δεν θα ε, απαιτήσει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, είναι όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο, μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση του νέου Επιτρόπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σφάμπ, έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας, ε, αλλά οι συγκεκριμένες ε, δεν αναφέρετε τι συγκεκριμένε προτάσει που θα ήθελα να δω να εφαρμόζονται καλύτερα στα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μου δώσετε παράδειγμα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που θα πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα. Στι γραπτές σα παρατηρήσει, λέτε ότι η πολιτική των καταναλωτών θα πρέπει να προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα και ότι στην ε, Ευρώπη θέλουμε να έχουμε μια πραγματική κουλτούρα του καταναλωτή και θα είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στου καταναλωτέ ότι είναι δύσκολο να πετύχουμε μια οριζόντια προσέγγιση εντός της ε, Κομισιόν ε, και γι' αυτό θα πρέπει να καθυστερήσουμε τα θέματα θέματα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να σπρώξετε την Επιτροπή και ω ε, εισηγητή για την ε, οδηγία για τη δικαιώματα του καταναλωτή ε, ομιλώ δεν θα ήταν χρήσιμο να έχουμε περισσότερη πλήρη εναρμόνιση ώστε οι καταναλωτέ να γνωρίζουν ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη διότι έτσι θα γνωρίζουν καλύτερα ότι μπορούν να απαιτήσουν να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του. Ναι, πράγματι. Ε, μίλησα για κάποιες ε, εκρεμείς προτάσεις ε, που θα δούμε σύντομα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Ήδη όμως έχουμε νομοθεσία που αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Εάν λοιπόν επιβεβαιώσετε την υποψηφιότητά μου τότε Ε, θα ε, επιμείνω στην καλύτερη εφαρμογή της ε, ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό ισχύει για, τις, για τον αθέμητο ανταγωνισμό, τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα πρέπει να κάνουμε επίσης περισσότερα όσον αφορά τις επιγραμμικές αγορές, τις αγορές στο διαδίκτυο. και ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, ε, θέματα ε, ουδετερότητας του διαδικτύου. Πρόκειται για τομείς στους οποίους θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Επίσης ε, τα δικαιώματα των επιβατών στα διάφορα μέσα μεταφοράς και είναι θέματα για τα οποία θα συνεργαστώ και με τους άλλους επιτρόπους για να εξετάσουμε τον αντίκτυπο στους καταναλωτές ε, και να περασπιστούμε τα συμφέροντα των καταναλωτών ε, κατά την εφαρμογή ε, των σχετικών νομοθετημάτων στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε τώρα στην κυρία Evelyn Γκέπχαρτ για τον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Ένα λεπτό για τις ερωτήσεις σου έχεις Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μίμητσα, μόλις είπατε Α, περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας. Sie sagten gerade in ihren einführenden... Είπατε στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις ε, ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών που δεν εφημάζονται, δεν επιβάλλονται, δεν υπάρχουν κιόλας. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται εδώ και καιρό με αυτό το θέμα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επιβολή της νομοθεσίας και την τήρησή της. Ένας από τους τρόπους είναι να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο συλλογικέ αγωγές και δεν μιλώ με το class action αμερικανικού τύπου, αλλά συλλογικές προσφυγές ευρωπαϊκού τύπου. Και θα με ενδιέφερε να μας πείτε πόσο πρόθυμος είστε να προχωρήσετε και να κάνετε προτάσεις και εδώ ε, για να κάνουμε επιτέλους μία πρόοδο και σε αυτό το τομέα. Ο οριστής επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέπχαρτ. που θέσετε αυτό το θέμα και πραγματικά ε, ε, απασχολεί ε, εδώ και καιρό. Και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι ένα πολύ θέμα και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις όλοι υπέρ των καταναλωτών στο ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Όντως για να δρέψουμε τους πλήρει καρπούς της ενιαίας αγοράς για να επιτρέψουμε στην ενιαία αγορά να λειτουργεί, να μπορεί ο κόσμος να κάνει αγορές διασυνοριακά, ε, θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε και να καθησυχάσουμε τους καταναλωτές, να εμπιστεύονται ότι μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες ε, της εσωτερικής αγοράς. Οι συλλογικές ε, αγωγές, οι προσφυγές μπορεί ενδεχομένως να είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Θα κατανοείτε σίγουρα ότι... Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δεν έχει ακόμα επίσημα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην προετοιμασία αυτού του θέματος εγώ δεν μετήχα. Οπότε το να αποφανθώ γι' αυτό θα ήταν για μένα πολύ δύσκολο, όσο και άστοχο να μπω σε λεπτομέρειες για την επερχόμενη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω όμως επίγνωση του θέματος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μου ενημερώθηκα ότι προσεχώς θα κατατεθεί πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα ασχολείται ε, με αυτά τα ζητήματα των συλλογικών αγωγών ή προσφυγών με έναν τρόπο ε, εγκάρσιο, συνολικό, συνεκτικό όπως άλλωστε ζήτησε και πρότεινε το Κοινοβούλιο σε έκθεσή του. Προσεχώς σε περίπτωση που επιβεβαιωθώ και διοριστώ, θα ασχοληθώ σε λεπτομέρειες και θα μελετήσω αυτά τα θέματα και με χαρά να ε, το προωθήσω για να δω σε ποιο βαθμό αντανακλά ε, πραγματικά τα συμφέροντα των καταναλωτών να έχουν την ευκαιρία συλλογικά να προσφεύγουν. Όχι σε διαδικασίες ε, ε, διακανονισμών και επίλυσης διαφορών και διαιτησίας ιδιαίτερα άσκοπων. Το θέμα δεν είναι θα έχουμε περισσότερες ή λιγότερες ε, δικαστικές αγωγές, αλλά ε, κατά πόσο θα έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές στην εσωτερική αγορά. Όντως το θεωρώ ασμήμα τμήμα της μελλοντική μου εργασίας και των ευθυνών αν αναλάβω. Εύελιν Κεπχάρτ. Συμπληρωματική επερώτηση. Ναι. Εγώ ρώτησα την προσωπική σας γνώμη. Ξέρω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ρώτησα αυτό. Ε, άλλο ρώτησα, εσείς προσωπικά τι φρονείτε. Σωστά κατάλαβα ότι ε, προσωπικά θα ήσασταν υπέρ μιας τέτοιας πρότασης να υιοθετηθεί. μάλιστα κύριε Γκέπχαρτ. Καταρχήν είμαι υπέρ ενός πλαισίου συλλογικών προσφυγών που θα σέβεται την εθνική νομοθεσία και την ένομη τάξη της κάθε χώρας, όσο και τις παραδόσεις και το νομικό πολιτισμό. Και θα αντανακλά το γνήσιο συμφέρον των καταναλωτών. Γι' αυτό θα αγωνιστώ. Σε περίπτωση που και μόλις έρθει η πρόταση ενώπιό σας και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω, δεν είμαι βέβαιος για το λεπτομερές περιεχόμενο της εν λόγω πρότασης. Όπως πάντα, αυτό που με ενδιαφέρει και για το οποίο θα αγωνιστώ είναι να ε, προασπίζεται το συμφέρον των καταναλωτών. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί κατά πόσο η πρόταση είναι αυτή που χρειάζονται οι καταναλωτές. Όταν έρθει η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον του Κοινοβουλίου να αντανακλά πλήρω τα συμφέροντα και τις προσδοκίε των καταναλωτών για την προστασία των συμφερόντων τους, των δικαιωμάτων τους και για την τόνωση της εμπιστοσύνη τους στην ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Φιλελεύθερη τώρα, ο ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, καλώ ήρθατε στις Βρυξέλλες. Εμ Εκ μέρους της ομάδας μας θα ήθελα να σας συγχαρώ για ε, τα σημαντικά αυτά θέματα ε, με τα οποία ασχολείστε και ε, ως δανός και εκπρόσωπος μιας μικρής χώρας μπορώ να σας πω ότι πιστεύω ότι η Βρυξέλλες είναι ε, το καλύτερο μέρος να βρίσκεται κανείς. Ε, όσον αφορά την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και στα πλαίσια της οδηγίας αυτής θέτει το θέμα της μη διάκρισης λόγω έδρας. Νομίζω ότι αυτό θα έχει ατυχές αποτέλεσμα διότι ε, αυτό θα σημάνει ε, υποχρέωση πώληση ε, εταιριών ακόμα και σε, από τις εταιρείε ακόμα και σε χώρες όπου δεν γνωρίζουν τους, καταναλωτικούς, τους κανόνες που αφορούν τους καταναλωτές. Πώς βλέπετε εσείς το θέμα αυτό της μη διάκρισης λόγω έδρας ή τόπου Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι η ενιαία αγορά συχνά είναι κατακερματισμένη λόγω κάποιων εμπορικών πρακτικών ε, και αυτό ισχύει και για τις αγορές στο διαδίκτυο ισχύει και όσον αφορά τις ε, αγορές που κάνει κανείς στην πατρίδα του ή στο εξωτερικό. Και σκοπεύουμε να εξετάσουμε τον, κατακαιρματισμό της αγοράς, να εξετάσουμε τις εκκρίσεις που γίνεται λόγω εθνικότητας, λόγω τόπου κατοικίας, λόγω χρήσης ε, συγκεκριμένου τρόπου πληρωμών, ε, για παράδειγμα ε, μέσω κάρτας που έχει εκδοθεί σε κάποια συγκεκριμένη χώρα ή τις αγορές με κινητό. Ο Επίτροπος για την καταναλωτική πολιτική θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, να συνεργαστεί με τον Επίτροπο Μπαρνιέ όσον αφορά το θέμα αυτό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των τρόπων πληρωμών. Στην ε, οδηγία περί παροχής υπηρεσιών ε, τίθεται το θέμα αυτό της ε, διάκρισης λόγω τόπου κατοικίας, αλλά υπάρχει και η ρήτρα που λέει ότι εκτός εάν κάτι τέτοιο αιτιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια. Δεν έχουμε όμως ε, κατευθυντήρες γραμμές ε, σχετικά με το τι θα μπορούσαν να θεωρηθούν, ε, τι θα μπορούσαν να θεωρηθεί αντικειμενικά κριτήρια. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να καθορίσουμε τους βάσιμους λόγους διάκρισης ή μη και είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Το σώμα των Επιτρόπων, ε, στο Σώμα των Επιτρόπων θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Ε, να ρωτήσω όμως ε, από την απάντησή σας καταλαβαίνω ότι θα τεθείτε στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο θέμα αυτό, διότι έχουμε πολλές τέτοιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ναι, πράγματι. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εσωτερική αγορά να ωφελεί τους καταναλωτές, να ωφελεί όμως και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, ε, έχουν πρόσβαση σε νομική εμπειρογνωμοσύνη, μπορούν να αναλύσουν προσεκτικά τους ε, κανόνες προστασίας, τους κανόνες ασφαλείας ε, στην αγορά. Αλλά με ίσους όρους ανταγωνισμού ε, όσον αφορά τους τρόπους πληρωμών κλπ. μπορούμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ριούλε. Αξιότιμη κύριε Μίμητσα. Χάρηκα πολύ για αυτό που είπατε και το καλωσορίζω ότι το δικαίωμα στην επιβολή της νομοθεσίας και την εφαρμογή θα είναι προτεραιότητά σας. Όταν κανείς αναφέρεται σε αυτά τα θέματα, πολύ σύντομα εμφανίζεται η υποπτία της αγοράς. Περιμένουμε εδώ και χρόνια τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιτέλους ήλθαν και το καλωσορίζουμε. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται πάρα πολύ ε, στο ρίσκο στην ανάλυση της, δηλαδή στους κινδύνους. Δυστυχώς όμως δεν το ορίζει αυτό. Τι εστί κίνδυνος ε, στην οδηγία. Και κάτι άλλο που βρίσκω ιδιαίτερα προβληματικό, η αρχή της προφύλαξης που μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ κεντρική, επίσης απουσιάζει από την οδηγία. Εσείς προτίθεστε να κάνετε βελτιώσεις, θα συνεργαστείτε μαζί μας προς την κατεύθυνση αυτή. Και να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Στα παιχνίδια κάθε χρόνο έχουμε το εξή φαινόμενο. Παραμονές Χριστουγέννων βγαίνουν σκάνδαλα. Ε, αυτό υπονομεύει βέβαια την εμπιστοσύνη των πολιτών στην υποπτία της αγοράς. Πώς μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε τους ελέγχους και να μην είναι μόνο μια ιστορία χριστουγεννιάτικη αυτή, αλλά με την καθημερινή δουλειά να αποτρέπονται τέτοια σκάνδαλα και σενάρια. Και επίσης θέλω να ρωτήσω κάτι για τις οριακές τιμές. Ε, μισό δευτερόλεπτο δικαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη Γερμανία για τα παιχνίδια, για τα βαρέα μέταλλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να κάνει βελτιώσεις εκεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μίμητσα. Κύριε Ρούλε, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όντως, είναι βασική ανησυχία αυτή των καταναλωτών, η ασφάλεια των προϊόντων και για τους ίδιους και για την υγεία τους. Θα σας έλεγα το εξής πραγματικά. Η ανάλυση κινδύνου αν εναρμονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα μας έδινε τη δυνατότητα να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Σε σύγκριση με την ανάλυση κινδύνου και την εκτίμηση από τις εκάστοτε εθνικές αρχές. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε, να οξύνουμε το πλαίσιο και τις οδηγίες, τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση και την εκτίμηση του κινδύνου. Και αυτό που χρειάζεται είναι πραγματικά να βελτιωθεί η συνεργασία ε, των αρχών που ελέγχουν την αγορά. Μεταξύ τους δηλαδή, με συνεργασία με βέλτιστες πρακτικές από τις οποίες θα μαθαίνουν όλοι και θα τις ε, διαδίδουν ε, στο δίκτυο εθνικών υποπτικών αρχών. Επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε και το βαθμό συνεργασίας με τη βιομηχανία και με τις... τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι αντιλαμβάνονται τη σημασία και την αποδοχή από πλευράς τους ότι χρειάζεται να παράγουν ασφαλή προϊόντα. Ε, αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν για την, ε, τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς αγγίζει πολλά τέτοια θέματα συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης της συνεργασίας και του συντονισμού σε επίπεδο κρατών μελών. Και υπάρχει πρόταση ε, να γίνει πιο συστηματική ανταλλαγή απόψεων και ο διάλογος ε, μεταξύ των εθνικών υποπτικών αρχών έτσι ώστε να είναι ασφαλή το περιβάλλον και ασφαλή τα προϊόντα. Ε, μπορώ να κάνω μια επερώτηση κυρία Ρούλε. Μα δεν απαντήσατε ακόμα συγκεκριμένα για το πώς ορίζεται τον κίνδυνο. Δεν θα πρέπει ανά την Ευρώπη να έχουμε κατακαιρματισμένους ε, ορισμούς, αλλά ενιαία αντιμετώπιση, αλλά και ένα ενιαίο ορισμό. Και κάτι άλλο που αναφέρατε είναι η ευθύνη της βιομηχανίας. Πώς θέλετε να συνδέσετε περισσότερο τη βιομηχανία στον έλεγχο των αγορών, γιατί ξέρουμε ότι είναι υψηλό το κόστος και χρειάζεται, δείτε εδώ, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ασφάλεια συμβαδίζει με την ασφάλεια. Η επιστήμη, οι επιστημονικές έρευνες και οι επιστημονικές συστάσεις είναι αυτό που χρειάζεται για τον εντοπισμό των κινδύνων. Εντοπισμός επιστημονικός των κινδύνων επί τη βάση επιστημονικών αποδείξεων για τα κινδύνους που απορρέουν από ορισμένα συστατικά ε, ή τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι συνδεδεμένα. Άρα λοιπόν η βελτίωση της αξιολόγησης κινδύνου σημαίνει βελτίωση ε, του του επιστημονικού αντικτύπου στα θέματα ασφάλειας και αυτό προσπαθούν να κάνουν οι Κομισιόν με τις υπηρεσίες, τους, με τις υπηρεσίες της. Ε, πρέπει δηλαδή να υπάρχουν συγκεκριμένες γραμμές για καλύτερο η αξιολόγηση κινδύνου που θα χρησιμοποιούνται και καλύτερα σε εθνικό επίπεδο από τις αρχές ε, Εθνικές Αρχές Εποπτείας. Αυτός είναι ο τρόπος για να προχωρήσουμε και θα ήμουν ευτυχής εάν επικυρωθώ να είμαι κομμάτι όλων αυτών των προσπαθειών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Μπίλε εξονόματος τη Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εξ ονόματος ε, της ομάδας μου θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για τη νέα σας θέση. Στις γραπτές σας απαντήσεις αναφέρετε ότι σκοπεύετε να προωθήσετε τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς προς τους καταναλωτές και ότι αυτή θα είναι μια από τις προτεραιότητές σας. Κάτι το οποίο πολύ με ευχαρίστησε. Τι συγκεκριμένα ωφέλη σκοπεύετε να προωθήσετε προς τους καταναλωτές, πώς και πότε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπίλαν. Όντως η ενιαία αγορά, όπως έχουμε επανελειμμένα πει, πρέπει να λειτουργεί για τους καταναλωτές. Υπάρχει η ενιαία πράξη που προωθήθηκε πολύ εδώ, σε αυτό το σώμα, και από συγκεκριμένη επιτροπή ακόμα και το όνομα ο τίτλος της ενιαίας πράξης προέρχεται από αυτήν εδώ την ε, Επιτροπή και η πολιτική του καταναλωτή και τα συμφέροντα του καταναλωτή αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη της εσωτερικής ε, αγοράς, της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό και προσβλέπω, ε, αναζητώ τις ευκαιρίες, οποτεδήποτε πρόκειται για ένα ε, μεγάλο θέμα το οποίο ε, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, όπως ε, το Europe, η Ευρώπη 2020, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, θα πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να αποκομίσουμε πολύ περισσότερα από ότι η απλή μακροοικονομική εικόνα ή και να ε, ε, εντάξουμε εκεί περισσότερες προοπτικές ε, από την προοπτική του καταναλωτή και της ενιαίας αγοράς. Η ενιαία πράξη ζητά, προβλέπει πολύ συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα σε διαφορετικούς τομείς στην καταναλωτική πολιτική ή μέτρα για τον καταναλωτή που είναι ένα κομμάτι όλων αυτών, αλλά και πάλι πρόκειται για μια οριζόντια πολιτική που μπορεί σαφώς να συμβάλλει πλήρως στην επιτυχία της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό και συγκεκριμένες δράσεις θα πρέπει να προωθηθούν και να εκτελεστούν ώστε να λειτουργήσει η αγορά για τον καταναλωτή και ο καταναλωτής να αποκτήσει κεντρική θέση στην ενιαία αγορά κύριος Μπίλαν, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Πώς θα εμπλέξετε τα κρατημέλη και τους βουλευτές να συμβάλλουν στην νέα αγορά, πώς θα συνεργαστείτε με τα κρατημέλη ώστε να εξασφαλίσετε ότι θα ε, βοηθηθείτε για τα δικαιώματα του καταναλωτή και η πολιτική σας θα διαδίδεται, θα γνωστοποιείται, ιδιαίτερα εν ώψη των ε, ευρωεκλογών του επόμενου έτους και ποιες συγκεκριμένες πολιτικές σκοπεύετε ε, να χρησιμοποιήσετε για την πρόθεση για να γνωστοποιηθεί η εργασία της Ένωσης για τη βοήθεια προς τον καταναλωτή. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ήδη τόνισα τη σημασία του συντονισμού όλων των ενδιαφερόμενων φορέων που είναι τμήμα ή που επηρεάζουν την επιτυχία ή την αποτυχία της καταναλωτικής πολιτικής. Η συνεργασία με τα κράτη-μέλη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της γενικότερης, της ευρύτερης συνεργασίας, οπότε δεν θα αφήσω προσπαθειών ώστε να είμαι σε διαρκή επαφή με τα κράτη-μέλη και τις αρχές τους τις αρχές εποπτείας της αγοράς, ε, τις αρχές ε, επιβολής των μέτρων, ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός. Θα έλεγα πως πρόκειται για μια πολιτική που θα πρέπει να είναι δραστήρια, θα πρέπει να είναι ενεργή, ενεργητική. Ε, δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι ότου τα κρατημέλη να ξεκινήσουν να μεταγράφουν ε, την Ευρωπαϊκή Οδηγία ή να περιμένουμε μέχρι ότου να αρχίσουν να σκέφτονται για τις καλύτερες μεθόδους συνεργασίας στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή, αλλά θα πρέπει ενεργά και δραστήρια να έχουμε τακτικές επαφές με τις εθνικές ε, αρχές και να μην αφήσουμε να δοθεί εντύπωση ότι κάτι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ κάποια άλλα πράγματα γίνονται μόνο στο επίπεδο των εθνικών αρχών. Αυτή η συνεργασία και ο συντονισμός είναι πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ και τελευταίο στο γύρο των συντονιστών ο κύριος Πάσκα ε, εξ ονόματος του ΕΦΔΙ. συγγνώμη, ξέχασα τον κύριο Ντε Γιόγκ. Και μετά ο κύριος Πάσκα, εγώ φταίω, ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Ντε Γιόγκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Μίμητσα, η Επιτροπή μας εδώ, ΙΜΚΟ, ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα καταναλωτών και ενδιαφέρεται πάρα πολύ να κρατήσει στα χέρια της ε, τα θέματα των καταναλωτών και των συντονισμών. Γιατί υπάρχουν και άλλες επιτροπές που έχουν τέτοιες ε, αρμοδιότητες. Εσείς θα είστε προσεχώς ένας νέος επίτροπος από μια μικρή χώρα και θα ε, κληθείτε απέναντι στα μεγάλα βάρη, τα βαρέα βάρη, Κρούς, Μπαρνιέ, Ρέντινγκ, να συντονίζετε ε, τα θέματα των καταναλωτών. Πώς θα το κάνετε αυτό. Ε, και όλη η νομοθεσία, έχουμε ομάδες εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει οι καταναλωτές να εκπροσωπούνται σωστά ε, υποβολή ε, νομοθετικών προτάσεων παραμένει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει οι καταναλωτές να εισακούονται. Είστε υπέρ ενός νομοθετικού αποτυπώματος που τα ακούμε εδώ και χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, θεωρείτε ότι οι καταναλωτές και οι οργανώσεις τους έχουν αρκετή επιρροή σε αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεγιόγκ για την ερώτησή σας. πραγματικά καταλαβαίνω το εξή. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μου για την ακρόαση προσπάθησα να συγκρατήσω τον αριθμό των επιτρόπων με τους οποίους θα πρέπει να συνεργάζομαι για να προωθώ τα θέματα των καταναλωτών. Παντού σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές και μάλιστα σε πολύ πρώιμο στάδιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας με μελέτες αντικτύπου βεβαίως και ε, με την κοινοβουλευτική συνομοθετική εργασία. Και είναι παρακαλώ 11 τον αριθμό οι επίτροποι ε, στο σώμα των επιτρόπων που με τον α β τρόπο ασχολούνται, επηρεάζουν ενδεχομένω τα θέματα των καταναλωτών και τα συμφέροντά τους στους τομείς πολιτικής. Η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο και περισσότερο εργάζεται εγκάρσια δεν υπάρχουν κάθετοι τομείς πολιτικής πυλώνες έτσι που να αφορούν ένα και μόνο επίτροπο. Είναι περισσότερο διάδραση, αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των πολιτικών. Και η πολιτική των καταναλωτών ε, γράφεται πάρα πολύ ωραία σε αυτό το πλαίσιο ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, ο δικός μου ρόλος και θα ήταν ε, να ε, είναι ε, τα συμφέροντα των καταναλωτών έμπρος στο βαρύ, δηλαδή από την αρχή, από το πρώιμο στάδιο της νομοθεσίας, αλλά και στην επιβολή στη συνέχεια. Τι εννοώ, για να μπορούν καλύτερα οι πολίτες να δέχονται και να κατανοούν και όλα τα υπόλοιπα αν τα δικά τους συμφέροντα από την αρχή συνυπολογίζονται και θα μπορούν καλύτερα να δέχονται ε, τις υπόλοιπες πολιτικές. Αυτό μας ενδιαφέρει, τα γνήσια πραγματικά συμφέροντα των καταναλωτών να αντανακλώνται και να προάγονται στην νομοθεσία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ακριβώς έτσι βλέπω το συντονισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Supplementary, συμπληρωματική ο κύριος De ε, Καλές οι προθέσεις, αλλά πολύ ασαφής η απάντηση. Ε, παράδειγμα, κοιτάξτε τα δικαιώματα των επιβατών. Ο κύριος Κάλλας είναι αρμόδιος, αλλά βλέπουμε και καταναλωτές που θέλουν να έχουν δικαίωμα ε, παντού, εξαρτήτως από το μέσο μεταφοράς. Αυτό είναι το δικαίωμα των καταναλωτών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβαίνει σε αποσπασματικές ρυθμίσεις κατακαιρματισμένες για συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς. Λοιπόν, εκεί θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να εισακούονται οι καταναλωτές και να επηρεάζουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για τη συμπληρωματική σας ερώτηση. Το έχω συζητήσει ήδη αυτό με τον Αντιπρόεδρο Κάλλας. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε, να ε, κάνουμε καλύτερη την ε, υφιστάμενη νομοθεσία για τα δικαιώματα των ε, επιβατών και συμφωνούμε εδώ για κοινέ προσπάθειες για τα συμφέροντα των καταναλωτών και πώς αυτά θα προάγονται στην κοινή μας προσπάθεια. Ακριβώς αυτό το τομέα λοιπόν τα δικαιώματα των καταναλωτών, των επιβατών με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Γιατί εγώ τρεις εβδομάδες είμαι στις Βρυξέλλες και η βαλίτσα μου ακόμα να έρθει. Ε, ούτε ξέρω που βρίσκεται, ούτε ξέρω τι να κάνω. <laughs> Με, με ενημέρωσαν για αυτή την ακρόαση, αλλά για το πού θα βρω τη βαλίτσα μου όχι. Ε, κάπου στο αεροδρόμιο των Βρυξελών είναι χαμένη. Βεβαίως χρειάζεται βελτίωση ε, των δικαιωμάτων των επιβατών για να βρουν τη βαλίτσα τους που δεν έχει χαθεί. Απλώς είναι σε ομοιρία κάπου. Εντάξει, καλές οι απεργίες και τα δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει να υπάρχουν και σαφείς διατάξεις για το ε, ποιος είναι υπεύθυνος και αρμόδιος όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα απώλειες και καθυστερήσεις ε, αποσκευών. Α, μάλιστα πρέπει να πείτε ότι έχει ίδιο συμφέρον. Ε, ο Επίτροπο εδώ το δηλώνει ο οριστής. Ο κύριος Πάσχα. Ευχαριστώ. E, Αγαπητέ ε, υποψήφι επίτροπε. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ σε εσά και στους πολίτες της Κροατίας η συμμετοχή, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σας προσφέρει ψηλότερη ποιότητα ζωής και καλύτερο μέλλον. Ε, τώρα, μία από τις αρμοδιότητές σας θα είναι να ενημερώνετε το κοινό για τα δικαιώματά του, τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους. Τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε σε αυτό το τομέα? Yes, thank you very much, first of all, for Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις καλές ευχές σας, για τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Πρόκειται για έναν στόχο τον οποίο επιδιώξαμε για πολλές δεκαετίες. Uh, και τώρα πια γίνεται πραγματικότητα. Βελτίωση της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών συμπεριλαμβανομένων των Κροατών πολιτών ε, Λίαν συντόμως, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό τμήμα της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής καταναλωτή. Εάν θέλουμε λοιπόν να βασιστούμε στους βασικούς πυλώνες αυτής της πολιτικής, οφείλουμε να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο ασφάλειας της αγοράς στο σημερινό, αλλά και να βελτιωθεί. Επίσης, χειραφέτηση των καταναλωτών και μεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά την επιβολή των νόμων και των προδιαγραφών. Φυσικά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε η ε, καταναλωτική πολιτική, να, η πολιτική μάλλον για τον καταναλωτή, να ενταχθεί σε όλες τις άλλες πολιτικές, όλες τις δραστηριότητες και τα μέτρα που προωθούν και ε, την εσωτερική αγορά και την καθιστούν μια πραγματικότητα. Για τα δικαιώματα του καταναλωτή, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να σας εξηγήσω πόσο θα ήθελα να προχωρήσω μαζί με την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ όσον αφορά τη βελτίωση του πλαισίου των ε, δικαιωμάτων του καταναλωτή και έπειτα έχω και ένα πολύ συγκεκριμένο έργο, αν επικυρωθώ, να είμαι υπεύθυνο δηλαδή για την εφαρμογή την επιβολή μάλλον των δικαιωμάτων του καταναλωτή και αυτό Αυτές θα είναι δράσεις που θα πρέπει συγκεκριμένα να αναλυφθούν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Πιστεύω πως μια γρήγορη ρύθμιση διαφορών είναι και αυτό το τμήμα των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Είστε έτοιμος να ενημερώσετε τους ε, πολίτες για έναν αποτελεσματικό και ταχύ τρόπο επίλυσης διαφορών. Ναι, βεβαίως. θα σκεφτούμε την ενημέρωση του καταναλωτή, όχι την υπερβολική ενημέρωση, δηλαδή την υπερφόρτωση με ένα σωρό πληροφορίε, αλλά μια ε, αποτελεσματική και ταχύα ενημέρωση έτσι ώστε να καθίστανται τα δικαιώματα κατανοητά. Ε, αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα της δράσης που θα αναλάβουμε και ως προς αυτό... Θα ήθελα να είμαι ένα σημαντικό κομμάτι των κοινών προσπαθειών που θα φέρουν την πολιτική του καταναλωτή στη, στα top των αποτελεσματικών μέτρων άσκησης πολιτικής. Ε, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και έτσι ολοκληρώνει το γύρο των ε, συντονιστών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές που ήταν πολύ πολύ ε, ε πειθαρχημένοι. Οι δικέ σα απαντήσει, ωστόσο ήταν ε, κάπω μακρύτερες κύριε Πίτροπε. Ίσως λοιπόν να ακούσετε πιο πολύ το σφυράκι καθώς θα προχωράμε γιατί διαφορετικά θα χάσουμε, θα μας λείπει χρόνο στο τέλος. Ε, να προχωρήσουμε στους άλλους πέντε ομιλητές από την Επιτροπή να σας θυμίσω. Γιουρά. Mr. Plenkovic ε, from Croatia, so we start with Mr. for one minute question. Ξεκινάμε με τον κύριο ε, Ζουβά. Κύριε Επίτροπε, και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας συγχαρώ για την ένταξη της όμορφης χώρας σας στην Ένωση. Θα ήθελα να συνεχίσω μετά από την ερώτηση της κυρίας Γκέμπαρντ σε σχέση με τις συλλογικές προσφυγές. Ε, το 2012 ε, το Ευρωκοινοβούλιο υποστήριξε τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος με την προϋπόθεση ασφαλιστικών δικλείδων. Το σύστημα αυτό είναι απαραίτητο γιατί οι καταναλωτές πρέπει να προστατευτούν διότι υπάρχουν εθνικές νομοθεσίες πολύ σκόρπιες και διαφορετικές αλλά το θέμα των ασφαλιστικών δικλείδων είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η κυρία Γκέμπαρντ σας ρώτησε, είστε υπέρ εσείς, εσείς και όχι η Κομισιόν γενικά, είπατε ναι, ναι, απαντήσατε ναι υπό δύο όρους. Και ο πρώτο όρο είναι να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του, τα συμφέροντα του καταναλωτή. Συμφωνώ με αυτή είναι η βασική αρχή. Και δεύτερο όρο είπατε υπό την προπόθεση ότι γίνεται σεβαστή η εθνική νομοθεσία και ομολογία. Επιτρέψατε μου να σας πω ότι εδώ διαρκώς τσακωνόμαστε με τις εθνικές νομολογίες και αν από την αρχή μας λέτε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το, την ε, ε, εθνική ε, νομοθεσία και νομολογία, θα έχουμε πρόβλημα. Το δικαίωμα για προσφυγή στα θέματα του περιβάλλοντος είναι δικαίωμα ή θα έχει να συγκρουστεί με την εθνική νομολογία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζουβά που, ήρθατε, που επανήλθατε στο θέμα της, εθνική, της ε, συλλογικής προσφυγής γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα αξιοπιστίας και πολιτικής για τον καταναλωτή εν γέννη. Και πάλι θα πρέπει να σας ζητήσω την κατανόηση να κατανοήσετε μάλλον ότι είναι πολύ δύσκολο για μένα να μπω σε λεπτομέρειες σε σχέση με τις προτάσεις που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και διατυπωθεί από την Κομισιόν. Αυτό που θα ήθελα να επαναλάβω ωστόσο είναι ναι, είμαι υπέρ και είμαι υπέρ εάν ε, και ε, επικυρωθώ εν γέννη για την συνεπή και οριζόντια προσέγγιση που θα λάβει υπόψη, θα ασχοληθεί με την προστασία του καταναλωτή, για με τον ανταγωνισμό, την προστασία του περιβάλλοντος, τις καλύτερες πρακτικές μέσα στην εθνική νομική παράδοση. Υπάρχουν ε, εθνικές νομικές παραδόσεις όσον αφορά τις συλλογικέ προσφυγές που δείχνουν ότι τα προβλήματα, τα υπερβολικά προβλήματα ε, και οι διαφορές ε, μπορούν να λυθούν μέσω αυτής της πρακτικής. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αντλήσουμε πείρα από τις εθνικές πρακτικές και αυτή να τη χρησιμοποιήσουμε για την πρωτοβουλία συλλογικής προσφυγής. Θα ήθελα επίσης να σας τονίσω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θα πρέπει να σεβαστούμε εν γέννη την ευρωπαϊκή νομική παράδοση και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε βήμα θα μας οδηγεί σε στέρεο έδαφος. Μπορεί να μην είναι αυτή η πρόταση που άμεσα θα αντιμετωπίσει όλες τις προσδοκίες και τα προβλήματα των καταναλωτών, αλλά με δουλειά θα, είναι πιο, θα γίνει πιο ρεαλιστική η πρόταση αυτή. Σα ευχαριστώ Επίτροπε. Μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Η παρατήρηση είναι ότι ο σεβασμός τη Εθνική Νομοθεσία είναι απαραίτητος. Ε, γι' αυτό συμφωνούμε. Απλά θα πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές χρησιμοποιείται ω άλοθη για να μην προχωρήσουμε. Ε, γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε αγαθοί. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ε, ε, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και ότι είναι τεχνικό το θέμα και ότι δεν μπορείτε τώρα να μπείτε στις λεπτομέρειες. Απλώς εμείς φοβόμαστε ε, όπως αυτό που ισχύει, αυτό που ισχύει στη ΣΥΠΑ, δηλαδή η αποζημίωση ως τιμωρία. Αυτό δεν το θέλουμε. Αυτό δεν το θέλουμε και θα ήθελα να ξέρω αν επί της ουσίας είστε μάλλον υπέρ ή κατά. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Again, you are definitely trying to get some, if not commitment. Προσπαθείτε να καταλήξετε σε κάποια δέσμευση ή εν πάση περιπτώσει πολύ συγκεκριμένη άποψη του υποψηφίου επιτρόπου για αυτό το πολύ λεπτό θέμα. Το θέμα όμως αυτό είναι λεπτό γιατί ακριβώς δεν υπήρχε δεν, δεν έχει υπάρξει ακρι, ακριβής οριοθέτηση και περιγραφή του θέματος. Ας, ε, έχω πάντως την εντύπωση ότι να συνεργαστούμε πρέπει να δουλέψουμε μαζί ώστε να να αποφύγουμε το θέμα των ποινών μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα συλλογικής προσφυγής. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, ως, εγώ μπορώ να το κάνω ως Επίτροπος για την προστασία του καταναλωτή και την πολιτική του καταναλωτή. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι ένα ε, σημαντικό τμήμα αυτής της διαδικασίας μαζί με όλους όσους τελικά θα σχηματίσουν αυτήν την, το περιεχόμενο της ε, έννοιας της συλλογική προσφυγής είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω, Επίτροπε Μιμίτσα. Καλωσορίσατε. ορίσατε. Τώρα, σύμφωνα με ε, έρευνες, η ικανοποίηση των καταναλωτών σε σχέση με την αγορά ενέργειας, την ενέργεια αφορά η ερώτησή μου, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι τιμές διαρκώς αυξάνονται και αυτή η τάση θα συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια. Γνωρίζουμε ότι η άμεση και η έμεση πρόσβαση συνδέεται με τα με του λογαριασμού των καταναλωτών και ότι το κόστος μεταφέρεται από τους μεγάλους στους μικρούς καταναλωτές και διαταράσσει την διαφάνεια της αγοράς καθώς και εκθέτει τα ευάλωτα νοικοκυριά. Η, ε, η αγορά η γενιά θα πρέπει να λειτουργεί προ όφελο των καταναλωτών. Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να υπάρξει διαφάνεια στι τιμέ και να απλοποιηθούν οι λογαριασμοί της ενέργειας. Τι μέτρα θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με τα κράτη-μέλη ώστε να προστατέψει τους ευάλωτες καταναλωτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που αναφέρατε αυτό το ερώτημα που πραγματικά έχει αντίκτυπο στην καθημερινή μας ζωή και ιδιαίτερα αυτό το καιρό. Για πολλούς καταναλωτές ε, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικό αέριο. Δύο διαδικασίες ε, είναι σε εξέλιξη στην αγορά ενέργειας. Η μία είναι η πορεία της αύξησης των τιμών για την ενέργεια, λόγω της αύξησης των τιμών ε, των καυσίμων, ε, των χαμηλών επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές, στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και άλλες απαιτήσει που στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν οι φορείς της αγοράς και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει πάντοτε να μεριμνούμε ώστε οι τιμές λιανικής για την ενέργεια να αντιστοιχούν στο κόστος της χονδρικής παραγωγής που αυξάνεται, ενώ το κόστος λιανικής δεν πρέπει να αυξηθεί πάνω από μια λογική αύξηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε το πακέτο για την ενέργεια. Και αυτό είναι μια διαδικασία ώστε η αγορά ενέργειας να γίνει πιο ανταγωνιστική ε, και πιο ελκυστική για τον καταναλωτή. Πρέπει να διερευνήσουμε τα πλήρη ανταγωνιστικά ωφέλη που μπορεί να προσφέρει το πλήρες πακέτο για την ενέργεια στους καταναλωτές. Ναι, η τιμολόγηση είναι ένας τομέας όπου ήδη έχουμε προβεί σε διάφορες δράσεις ώστε να δημιουργήσουμε ένα πιο μια πιο καθολική διαδικασία τιμολόγηση, ιδιαίτερα τη ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους καταναλωτέ, και αυτό ήταν και τμήμα του εγχειρήματο ε, πίνακα επιδόσεων και των ε, πορισμάτων αυτού. Με βάση περιπτώσει, η Κομισιόν με τις υπηρεσίες της ενέργειας από κοινού θα ξεκινήσουμε σύντομα μια μελέτη, μελέτη για τους τους καταναλωτές σε διάφορα τμήματα της αγοράς, ιδιαίτερα στην ενέργεια. Ευχαριστώ, αλλά υπάρχουν και οι ρυθμιστικέ αρχέ και θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι ο ρόλο που πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουν οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ αφενό και επίση η ε, ρυθμιστική αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΣΕΡ στην προσπάθεια ενοποίησης αυτής της αγοράς, πώς μπορούν να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες αυτών των ρυθμιστικών αρχών προς όφελος των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ. Οι αρμοδιότητες αυτών των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενισχύονται με το τρίτο πακέτο για την ενέργεια. πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή και να έχουν πρόσβαση σε περισσότερους χώρους για να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν με τις ρυθμιστικές τους δραστηριότητες περισσότερους καταναλωτές. Έτσι δηλαδή όχι απλώς να λαμβάνουν υπόψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές και τις, τα κριτήρια ή τις υποχρεώσεις των παραγωγών, αλλά ταυτόχρονα να ε, θέσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών στο επίκεντρο της πολιτικής για την ε, αγορά της ενέργειας, διασφαλίζοντα τη δυνατότητα του καταναλωτή να συγκρίνει και να επιλέγει. Αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ μπορούν να συμβάλλουν. Η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή, από την πλευρά τη, χρειάζεται περισσότερου πόρου για να είναι πιο αποτελεσματική και να παρακολουθεί αν υπάρχει πραγματικό ανταγωνισμό στην αγορά και να ε, ελέγξει κατά πόσον ε, υπάρχουν στερευλώσεις στην αγορά ή η μείωση του ανταγωνισμού. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τένκοβιτς είναι ο επόμενος ε, ομιλητής. Θα ήθελα να ζητήσω να υπάρχει ησυχία. Ο κύριος Τένκοβιτς, Πλένκοβιτς από την Κροατία. Σας ευχαριστώ κύριε Χάρμπορ και καλωσορίζω τον κύριο Μίμητσα. Φυσικά θα μιλήσω στα προωτικά. Έχω ένα γενικό ερώτημα για να αντιληφθώ καλύτερα την άποψή σας σε σχέση με τις τάσεις που αναπτύσσονται στο πολιτική ε, προστασία του καταναλωτή. Η φιλοσοφία των προηγούμενων επιτρόπων ήταν να δοθεί μεγαλύτερη εξουσία στον ε, καταναλωτή, να αποκτήσει ο καταναλωτής μεγαλύτερες ε, δυνατότητες. Και η άποψη που θα ήθελα να γνωρίζω η δικιά σας είναι χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερα εργαλεία οι καταναλωτές έτσι ώστε να αποκτήσουν καταναλωτική συνείδηση και να βρίσκονται σε θέση να προστατεύσουν τα δικαιώματα τους καλύτερα. θα αξιοποιήσω τη δυνατότητα που έχω να μιλήσω στα κροατικά, Μια και με ρωτήσατε στα κροατικά. Πράγματι, για να αποκτήσει ένας καταναλωτής μεγαλύτερη δύναμη, χρειάζεται να αναλυφθούν πολιτικές ε, προστασίας του καταναλωτή και αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Μιλούσα λοιπόν για την Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον καταναλωτή, εκεί ορίζονται οι βασικές δραστηριότητες που πρέπει να αναλάβουμε, βασικές δράσεις. Μετά την ασφάλεια που ήταν ο πρώτος πυλώνας της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον καταναλωτή, ο δεύτερος πυλώνας, και αυτό δεν είναι τυχαίο, συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση της θέσης του καταναλωτή στην εσωτερική, στην ενιαία αγορά. όπως έχω πήγε στο παρελθόν, θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να προωθήσω αυτές, αυτή την ατζέντα. Που σημαίνει επίσης ότι θα χρειαστεί να αναλυθούν νέες πολιτικές ή να μεταβληθούν οι υφιστάμενες με στόχο την ε, ενημέρωση των καταναλωτών έτσι ώστε να αποκτήσουν συνείδηση να αντιληφθούν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που παίζουν στην εσωτερική αγορά και πόσο έχουν στα χέρια τους την δύναμη να μεταβάλουν τις πολιτικές που ακολουθούνται και με τις οποίες ευελπιστούμε να ε, ξεκινήσει η ανάπτυξη. Εάν δεν δουλευτούν οι ίδιοι οι καταναλωτές δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Οι καταναλωτές έχουν τη δύναμη στα χέρια τους, την οικονομική δύναμη και θα πρέπει να έχουν και τα νομικά βοηθήματα που ε, χρειάζονται για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Χωρίς αυτή την συνειδητοποίηση δεν μπορούμε να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση της εσωτερικής αγοράς. Και αντιλαμβάνομαι το ρόλο μου ως ένας άνθρωπος που θα θέτει τους καταναλωτές στο επίκεντρο οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη. Σε ευχαριστώ για την απάντησή σας. Εσείς πώς ορίζετε εκείνη την ομάδα στην οποία αναφερόμαστε με τον όρο ευάλωτοι καταναλωτές. Ποιοι θα ήταν αυτοί. Είναι ένας καταναλωτής ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς τα δικαιώματά του, είναι ένας ε, καταναλωτής που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, είναι ένα άτομο με αναπηρία ή κάποιος ε, ο οποίος ε, για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί ποια είναι τα δικαιώματα του ως καταναλωτής ότι βρίσκεται σε κάποια μειονεκτική θέση. Πώς εσείς ορίζετε λοιπόν την έννοια του ευάλωτου καταναλωτή. στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τους ε, καταναλωτές αναφέρονται δύο προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Μία από αυτές είναι η βιώσιμη κατανάλωση και η δεύτερη είναι το ζήτημα των ευάλωτων καταναλωτών. Δηλαδή εκείνων που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, αυτή η έννοια του ευάλωτου καταναλωτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να οριστεί όχι μόνο ανάλογα με την προσωπική άποψη του καθενός, αλλά και με τεχνικά κριτήρια όσο το δυνατόν πιο ε, ολιστικά, ε, ε, συνολικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει την εκπόνηση μιας μελέτης με στόχο να καθορίσει ποια είναι τα στοιχεία που καθιστούν έναν καταναλωτή ευάλωτο σε διάφορους ε, τομείς της αγοράς, την ψηφιακή αγορά, την αγορά ενέργειας κτλ. Νομίζω ότι έτσι με αυτή τη μελέτη θα έχουμε στα χέρια μας ε, μια βάση συζήτησης για να ε, επιλέξουμε τα μέτρα που χρειάζονται για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Η κυρία Σάντελ Μόζε, καλώς ορίσατε. Έχω δύο ερωτήσεις για σας. Πρώτον, θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο να αναφέρεται η αρχή της προφύλαξης στον κανονισμό. Και δεύτερον, σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, την υλοποίησή τους. Γνωρίζουμε ότι πολλά κράτη-μέλη δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Εσείς προσωπικά θα επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπουργούς, με τους αρμόδιους στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να τους παροτρύνετε να υλοποιούν και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ως συνήθως οι εύκολες ερωτήσεις είναι και πιο δύσκολες να απαντηθούν. Αυτή τη φορά δεν με τροβάξατε και πολύ. Όσον αφορά την Υλοποιεί την εφαρμογή όλες τις ε, νομοθεσίες προστασία του καταναλωτή, θα προσπαθώ να προλαμβάνω καταστάσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Και πάλι να αναφέρω ότι αυτό είναι ένας από τους πυλώνες της ατζέντα για τους καταναλωτές. Για να απαντήσω ευθέω, ναι, θα ε, έχω τακτικές συναντήσεις και τακτικές επαφές με τους αρμόδιους υπουργού και τις αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη προκειμένου να γνωρίζω και τις δικές τους απόψεις, τις δικιά τους, τα, δικα, τα, τα προβλήματα που εκείνες έχουν, εκείνοι και εκείνες έχουν εντοπίσει στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και επίσης για να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις, την εμπειρογνωμοσύνη που αποκτάται σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της ε, παρακολούθησης της αγοράς. Το πακέτο για την ε, μέτρων για τα παρακολούθηση της αγοράς που ε, συζητείται με το θέτη. θεωρώ ότι είναι μια επιπλέον δράση με στόχο την βελτίωση των δράσεων που ήδη αναλαμβάνουν οι εθνικές αρχές. Δηλαδή δίνει στις εθνικές αρχές και νέα εργαλεία και νέες δυνατότητες, για παράδειγμα απροειδοποίητους ελέγχους, επιτόπου στους, ε, στόπους παραγωγής προϊόντων, μπορούν επίσης να ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες, να προσάγουν στη δικαιοσύνη παραγωγού οι οποίοι δεν ε, εφαρμόζουν τις, τον κανονισμό. Αυτές λοιπόν οι δραστηριότητες δεν θα μπορούσαν να αναλυφθούν χωρίς να υπάρχει και μια συνεισφορά από ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Μιλτρία, αλλά δεν απαντήσατε στην πρώτη μου ερώτηση, δηλαδή εάν συμφωνείτε με ότι θα πρέπει να αναφερθεί η αρχή της προφύλαξης ευθέως και ρητά μέσα στον κανονισμό, κάτι που πιστεύω ότι είναι απαραίτητο. Κύριε Μιμίτσα, εάν επιβεβαιωθώ, θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας για να το συζητήσουμε, για να υπάρξει διάλογος και να βρεθεί η βέλτιστη συνδυαστική λύση ε, σε συνεργασία με τους ε, βουλευτές, τους ευρωβουλευτές αυτής της Επιτροπής και όλων τους άλλους σε οποιαδήποτε πρόταση υποβάλλει η Επιτροπή. Θα εξετάσω εντελεχώς όλες τις προτάσεις και οποτεδήποτε υπάρχει δυνατότητα να επιτύχουμε κοινού συμβιβασμού ή οποτεδήποτε η πρόταση που έρχεται από εσά, για παράδειγμα εδώ θα βοηθήσει ο κανονισμός να γίνει καλύτερος, να δώσει περισσότερες δυνατότητες για παράδειγμα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχέ, τότε ναι βεβαίω θα συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ κυρία Τούνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Οριστέντα Επίτροπε, ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι θέλετε να ενισχύσετε το επιγραμμικό εμπόριο. Ε, σας έγινε ερώτηση εάν προτίθεστε να επιταχύνετε το θέμα των συλλογικών αγωγών ε, προσφυγών και τώρα μας λέτε ότι το ταμείο είναι μείον και ότι ε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σωστά αυτό το μέσο των συλλογικών αγωγών στο διαδικτυακό εμπόριο. Μα γνωρίζετε ότι αυτό δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές, αφορά και τις επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους συναδέλφους της δικής μας Επιτροπής, διότι ε, ε, είμαστε πάρα πολύ στρατευμένοι σε αυτή την υπόθεση. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαμε επανειλημμένα συζητήσεις σχετικές και ε, ακούσαμε ότι αυτό μας κοστίζει ένα εκατομμύριο το χρόνο, τώρα ακόμα 8 εκατομμύρια. Έχουμε παραπλανήσει τους καταναλωτές οι οποίοι περιμένουν από εμά να δράσουμε. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά θα γίνει και δικό σας πρόβλημα. Λοιπόν, ε, συγκεκριμένα, πώς προτίθεστε να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Thank you very much, Mrs. for... Ευχαριστώ πολύ κυρία Τούν. Για λόγους χρονικούς ε, δεν απάντησα στο θέμα της ε, εναλλακτικής επίλυσης ε, διαφορών σε προηγούμενη ερώτηση. Γνωρίζω ότι εσείς ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για αυτό το θέμα και περίμενα ότι θα με ρωτούσατε κάτι τέτοιο και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, όντως, πλατφόρμες και μηχανισμοί για αυτή την επίλυση επιγραμμικών διαφορών είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα πρέπει και θα αποτελέσει ένα σημαντικό ε, τμήμα του χαρτοφυλακίου αυτού. Τώρα δεν έχουμε αρκετό χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες ή να αναλύσουμε το συνολικό πλαίσιο της αναλλακτική επίλυσης διαφορών. Μέχρι να γίνει αυτό λειτουργικό θα χρειαστούν 1,5 χρόνους και 2 και θα πρέπει να υπάρχει πλατφόρμα ODIR, ε, ODR που να υπάρχει σε όλες τις γλώσσες για την επιγραμμική επίλυση διαφορών και αυτό χρειάζεται χρηματοδότηση. Ε, θα έλεγα ότι σήμερα δεν είναι σαφής η εικόνα ούτε το τοπίο ότι ε, στο πρόγραμμα των καταναλωτών μπορούν να ικανοποιηθούν οικονομικά όλα τα αιτήματα και να λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα αποτελεσματικά. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την πλατφόρμα ODR. Κάνουμε όμως κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσουμε ε, το οικονομικό κόστος και την επιβάρυνση ε, για να λειτουργεί σε όλες τις γλώσσες. Είναι θέμα μετάφρασης αυτό. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να αντλήσουμε αυτά τα κονδύλια ε, ε, είτε από το πρόγραμμα των καταναλωτών είτε από άλλα προγράμματα για να ε, καλύψουμε το κόστος της μετάφρασης από ανθρώπους που πρέπει να γίνει αυτή, δεν που γίνεται ηλεκτρονικά. Καταλαβαίνετε ότι προσβλέπουμε στην κατανόηση και τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Μιμιτσά για την απάντηση αυτή. Αλλά καμιά ημερομηνία θα μας πείτε. Πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Μας ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Ε, μας είπατε ότι σκοπεύετε να μειώσετε το κόστος λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών. Ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά Υπάρχει ε, το ECC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών, που καμιά φορά επικαλύπτει την εργασία άλλων ε, συστημάτων, άλλες πλατφόρμες, γιατί βρίσκονται και σε δύο διαφορετικές γενικές διευθύνσεις. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να συντονιστούν. Το είπατε κι εσείς, ο Ευρωπαίος καταναλωτής μπερδεύεται ε, παίρνει άλλες προφορίες από διαφορετικές πηγές και τον οδηγούν σε σύγχυση όλα αυτά. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζει σε άλλο πλανήτη από τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε για όλα αυτά. Thank you very much for supplementary Σας ευχαριστώ πολύ για την επερώτηση αυτή, η οποία μπαίνει και σε λεπτομέρειες χρηματοδότηση πλατφόρμας ODR για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Εγώ μπορώ να δεσμευτώ ως προς τα εξή για την ίδια τη λειτουργία και ε, τη διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας αυτής ODR σε όλες τις γλώσσες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουμε και να το υλοποιήσουμε όλες οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα να δεσμευτώ για ένα χρονικό ορίζοντα αυτό θα εξαρθεί από τις χρηματοδοτικές πηγές και τα προγράμματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Με τον ΑΒ τρόπο θα πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη ε, προσπάθεια και μέχρι το 2014 το πλαίσιο που είχε αναφερθεί στην ατζέντα των καταναλωτών νομίζω ε, ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρήσουμε αυτή την ε, προθεσμία. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος γύρος ερωτήσεων ε, έληξε από την Επιτροπή ε, την ΙΜΚΟ και καλωσορίζω την κυρία Κρίστα Κλάς που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, περιβάλλοντος και θα κάνει και ερωτήσεις. Της παραδίδω την Προεδρία αλλά το χρόνο θα τον τηρώ εγώ. Έτσι μην νομίζετε ότι θα τη γλιτώσετε. Ε, η κυρία Κλάς, ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφοι ε, Χάρμπορη, Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, κύριε Μίμητσα, κύριε Οριστέντα Επίτροπε. Είναι μια επιτροπή επίσης που ασχολείται πάρα πολύ και ενέχεται με αυτά τα θέματα του δικού σας ε, χαρτοφυλακίου, περιβάλλον, ασφάλεια τροφίμων, προστασία καταναλωτών. Γι' αυτό σας καλωσορίζουμε και εμείς και είμαστε παρόντες. Στην περασμένη ερώτηση και στον περασμένο γύρο ερωτήσεων είδαμε πόσο εγκάρσιο, πόσο οριζόντιο είναι αυτό το θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Και στις επιτροπές λοιπόν του Κοινοβουλίου υπάρχουν αντίστοιχες αρμοδιότητες και μας αφορούν και τα δικά σας θέματα ε, τεχνολογικά, ιατρικά προϊόντα, ασφάλεια προϊόντων, καλλιντικά, ορισμένα χημικά και άλλα θέματα καταναλωτών. Είναι ζητήματα που αφορούν ε, και συμμετέχει η Επιτροπή μας και με μεγάλο προσωπικό και με μεγάλο ενδιαφέρον και με μεγάλη κινητοποίηση και, και θα έχουμε να πούμε και εμείς το λόγο μας ο οποίος θα βαρύνει και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συμμετέχουμε αναλόγως και αντιστοίχως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε διαπιστώσει ότι σε πολλά θέματα ε, συνεργαζόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε άρα ε, ποντάρουμε σε πολύ καλή συνεργασία με τον αρμόδιο επίτροπο. Έχουμε τρεις ομιλητές μόνο ε, από την Επιτροπή μας σήμερα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζέμπερ, μετά στην κυρία Μέρεντ και μετά στον Πέτερ Λίζε. Α, τώρα μου λέγουν ότι θέλει πρώτα ο Πέτερ Λίζε. Εντάξει, ο Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Οριστέντα Επίτροπε θα ήθελα να αναφέρω δύο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες ε, που είμαστε εμείς καθήλυνα αρμόδιοι και συνεργαζόμαστε αγαστά με την ΙΜΚΟ. Αυτό είναι τα ιατρικά προϊόντα και ε, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Χρειαζόμαστε καλύτερη προστασία των ασθενών αλλά και καινοτομία εμπροκειμένου. Οπότε σας ερωτώ συγκεκριμένα τι θα κάνετε για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Μένετε στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν προβλέπει προέγκριση είτε εθνική είτε ευρωπαϊκή. Θέλετε να δώσετε αλλού το κέντρο βάρους. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ε, προτάσεις για τι διαγνωστικές μεθόδους ε, που θέλουν να ενισχύσουν κάποιες προτάσεις τις οποίες δεν συμπεριλαμβάνει το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς ως οριστής επίτροπος πώς τα αξιολογείτε όλα αυτά. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Thank you very much, Dr. Ευχαριστώ πολύ, Dr. Λίζα. Όντως, συμφωνώ και προσβλέπω με χαρά να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος σε πολλά ε, ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την ασφάλεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των διαγνωστικών, των καλλιντικών και τα περιβαλλοντικά. Ε, αηφόρος, κατανάλωση επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα μπορούσα να σας παραθέσω και άλλους ε, τομείς και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ε, επανέρχομαι στην πρόταση για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που είναι ε, ενώπιον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αυτόν τον καιρό. Πρέπει να σας πω ότι θα είμαι πολύ ειλικρινής αν διοριστώ για να βελτιώσω μαζί σας στη συνεργασία όλα τα στοιχεία ασφάλειας στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, σε ό,τι αφορά την προέγκριση, πριν την κυκλοφορία στην αγορά δηλαδή, ε, όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ενίσχυση του υφισταμένου συστήματος των ε, οργανισμών που είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν και υπάρχει και ένα πολύ αυστηρό σύστημα επηρεασμού όσο και επαλήθευσης σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων των εθνικών αρχών όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού κινδύνου. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιλαμβάνει αλλαγή στη φιλοσοφία ή στην ε, προσέγγιση ως προς την προέγκριση ε, πριν την κυκλοφορία στην αγορά ε, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλού κινδύνου από ένα κεντρικό φορέα. Διότι εξ όσων γνωρίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διατηρήσει την τεχνολογία και την καινοτομία που είναι στην αιχμή του δόρατος αυτός ο κλάδος και αυτά τα προϊόντα στην Ευρώπη. Και ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε γι' αυτό και θα συνεργαστούμε Κατά τη διάρκεια της παρούσα κρόση, θα έχουμε σίγουρα και μεγαλύτερες και περισσότερες ευκαιρίες να μπούμε σε αυτό το θέμα της πρότασης για τα τεχνολογικά προϊόντα. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση ο κύριος Λίζερ. Ναι, μήπως συγκεκριμένα να μου απαντούσατε στις ερωτήσεις και στις δύο. <laughs> Εάν διοριστείτε και αναλάβετε το χαρτοφυλάκιο θα διατηρήσετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως έχει ή θα την αλλάξετε. Και τι λέτε για τις τροπολογίες για την ενημέρωση, το informed consent, ε, τη συνένεση κατόπιν ενημέρωση με τα λόγου γνώσεως. Ε, ο κύριος Μίμητσα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η παρούσα πρόταση για την διάγνωση in vitro ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ασφάλεια των ε, ε, γενετικών δοκιμών και των αντιστοίχων μεθόδων. Εγώ πώς βλέπω το ρόλο μου στην έγκριση αυτών των προτάσεων. Θα δεσμευτώ σε ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση με όλους ε, όσοι έχουν καλές προτάσεις και καλές πρωτοβουλίες και τροπολογίες για να αυξηθεί η ασφάλεια. Αλλά όχι μόνο η ασφάλεια. Αν διαπιστώσω ότι υπάρχουν καλές προτάσεις που επίσης ε, μετοπίζουν και τα δεοντολογικά ζητήματα και ζητήματα ηθικής χρήσης τέτοιων προϊόντων για γενετικές δοκιμές. Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ για να ενισχυθεί η ε, συνένεση ε, των ε, ενδιαφερομένων. Δηλαδή να ενημερώνεται σωστά ενδιαφερόμενος και να ε, ερμηνεύεται σωστά το αποτέλεσμα της γενετικής δοκιμής, να τα γνωρίζουν αυτά οι ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ, η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Κύριε Πίτροπε, εγώ ίσως να τα σας πω κάπως διαφορετικά, από διαφορετική γωνία από ότι ο κύριος Λίζε, αλλά πάντως θέλω απάντηση από σας. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Συμφωνείτε μαζί μου ότι η πρόταση της Επιτροπής για το ε, ιατροτεχνολογικό ε, προϊόντα και όχι για την in διάγνωση, Πάντως ε, δεν είναι απόλυτα σαφής για, τους, ε, για τα προϊόντα υψηλού κινδύνου. Δεν βελτιώνει δηλαδή την ασφάλεια των ε, ασθενών. Δηλαδή οι κοινοποιημένοι οργανισμοί εάν δεν ενισχυθούν οι δυνατότητές τους και οι γνώσεις τους δεν αρκούν για την ασφάλεια του ασθενή, πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη νομοθεσία, διαδικασία για το τεχνολογικό προϊόντα που μπορεί να περιλαμβάνουν, να περιέχουν μάλλον ενεργά δραστήρια τελικά. Είστε έτοιμοι να, είστε έτοιμοι να το υποστηρίξετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ροτ Μπέρεντ. Για αυτό το θέμα που μας φέρνει και πάλι στο, στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλού κινδύνου. Ίσως να είναι κάπως ε, λεπτό αυτή τη στιγμή να σχολιάσω την πρόταση της Κομισιόν, αλλά θα το κάνω έτσι Ελπίζω με τον κατάλληλο τρόπο. Ελπίζω ότι όταν οι συνομοθέτες, σε αυτή την περίπτωση οι ευρωβουλευτές, ε, καταφθάνουν με σωστά επιχειρήματα, σωστές τροπολογίες, βιώσιμες προτάσεις ώστε να ενισχυθεί το σύστημα της πρόσβαση στην αγορά για τα προϊόντα υψηλού κινδύνου, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια, εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω και να προσπαθήσω να βρω την καλύτερη δυνατή λύση, άσχετα ποια είναι η αρχική πρόταση της Κομισιόν. Πάντοτε μπορούμε να επανέλθουμε στην Κομισιόν, εφόσον συμφωνήσουμε ε, επί της ουσία η ουσία αυτή θα είναι το να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μας στους ε, οργανισμούς κοινοποίηση. Να, είμαστε, να, να υπάρχει ένας αριθμός ε, πυρογνωμών υψηλού επίπεδου, μπορεί να είναι και μικρός αριθμός των ε, οργάνων κοινοποίησης, δεν χρειάζεται να υπάρχουν τόσο πολλοί. Αλλά πάντως πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, ενισχυμένη εμπιστοσύνη σε αυτά τα σώματα και να αναπτυχθεί και μια επαλήθευση, μια δεύτερη ματιά από τις εθνικές αρχές. Όποιο σύστημα συνδυασμένων προσπαθειών μπορεί να ανεβρεθεί, θα προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε. Εγώ δεν θα ήθελα να επεκταθώ ιδιαίτερα όσον αφορά μια πλήρη μετακίνηση στην προς μια κεντρική έγκριση ή αδειοδότηση πριν από την κυκλοφορία στην αγορά, θα έμενα περισσότερο στον τομέα της, ε, ε, ε, ε εξασφάλισης των δραστηριοτήτων των κοινοποιημένων οργανισμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ που μένετε. Μάλλον εκτιμώ το ότι θέλετε να μένετε πιστό στην πρόταση της Κομισιόν. Μπορείτε όμως να, ωστόσο, να με διαβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να υπάρχει μια ε, άδεια για την κυκλοφορία στην αγορά των προϊόντων υψηλού κινδύνου, όποια και αν θα είναι αυτή η διαφορά. Ναι, σας ευχαριστώ. Φαίνεται πως, μου φαίνεται ότι η πρόταση της Επιτροπής ήδη τονίζει και αυτή τη διαφορά εισάγοντας επαληθεύσεις, ε, μάλλον διαδικασία επαλήθευσης ε, των ε, ιατρικών αρχών όπου αυτό είναι απαραίτητο πέρα από την έγκριση του οργανισμού κοινοποίησης. Υπάρχει δηλαδή αυτή η διάκριση που ήδη γίνεται ή μάλλον η επιπρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη εφόσον υπάρχει ανάγκη επαλήθευσης για τα προϊόντα υψηλού κινδύνου. Αλλά αν αρκεί, αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε από κοινού. Ευχαριστώ. Ρίχαρτ Ζέμπερ, από πλευρά μας. Ευχαριστώ. Ω Αυστριακό χαίρομαι ιδιαίτερα που ε, προσήλθε και η Κροατία στην οικογένειά μας. Ε, έχετε ένα χαρτοφυλάκιο πολύπλοκο και πολυδιάστατο και για τα καλλιντικά είστε αρμόδιος και γνωρίζετε ότι 70 δισεκατομμύρια ευρώ έχει ο κλάδος αυτός τζίρο το χρόνο και ε, χιλιάδες εργαζομένους ε, και καλύπτει το μισό της παγκόσμιας αγοράς. Έχουμε όμως και μια φιλόδοξη νομοθεσία για την προστασία των ζώων και στις 8 Μαρτίου απαγορεύτηκαν πλήρως στην Ένωση τα πειράματα σε ζώα ε, για τα καλλιντικά. Ε, γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει ένα παραθυράκι ακόμα αν χρησιμοποιούνται σε άλλα προϊόντα αυτά τα ε, οι ουσίες, όχι σε καλλιντικά δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα ακόμα να χρησιμοποιούνται πειραματόζωα. Και η δυσκολία είναι εδώ η διαχωριστική γραμμή και τα κράτη-μέλη παίζουν σπουδαίο ρόλο. Απαντώντας στον κύριο Σφαμπ προηγουμένως είπατε ότι Καμιά φορά το λιγότερο ε, σημαίνει περισσότερο. Αλλά εσείς πώς φαντάζεστε τον ηγετικό σας ρόλο ως επίτροπος, ε, να, πώς θα επιβάλλετε αυτή τη λεπτή διαχωριστική γραμμή. Ε, Ευχαριστώ κύριε Ζέμπερ. Όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα, τα πειράματα στα ζώα για την ανάπτυξη η απαγόρευση αυτών των πειραμάτων τηρείται από το Μάρτιο του 2013 και μετά και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Κάτι που το καλωσορίζω και είμαι ευτυχής που συνέβη αυτό πριν να αναλάβω το χαρτοφυλάκιο αυτό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας στην Επιτροπή. Ας δούμε λοιπόν όλες τις πτυχές της πλήρους ε, τήρησης και ε, εφαρμογής αυτής της απαγόρευσης. Πρέπει πολλά πράγματα να κάνουν οι εθνικές αρχές. Πρέπει να αναπτύξουν ένα πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών για να εξασφαλίσουν ότι τα πειράματα σε ζώα θα απαγορεύονται και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που ε, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πρόβλημα είναι όταν γίνονται πειράματα σε ζώα όχι για την δοκιμή των ε, συστατικών των καλλιτικών αλλά για την δοκιμή άλλων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται γενικότερα στη βιομηχανία ή σε άλλες αγορές. Εδώ είναι ζήτημα ερμηνείας της νομοθεσίας. Με χαρά θα παρακολουθήσω τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Για να δω. Ποια θα είναι η τελική ερμηνεία της νομοθεσίας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή και το βαθμό στον οποίο απαγορεύτηκαν οι δοκιμές στα ζώα. Η δική μου συνεισφορά δεν μπορεί να ξεκινήσει παρά μόνο μετά από περισσότερη μελέτη. Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες. Ναι, εγώ θα ενδιαφερόμουν για μερικά κριτήρια προσωπικά σας. Ε, τι θα θέλατε να δείτε. Εν περιπτώσει, έχω άλλη συγκεκριμένη ερώτηση. Το άρθρο 20 ε, ε, ισχυρισμοί προϊόντων. Άρθρο 20 του κανονισμού για τα καλλιντικά. Το είπατε. Θέλετε να αποφύγετε την παραπλάνηση των καταναλωτών. Αυτό πώς το βλέπετε. Yes, thank you for... Ε, Σας ευχαριστώ που θέτετε αυτό το θέμα των ισχυρισμών των προϊόντων ιδίως στον τομέα των καλλιντικών. Μια, ένας από τους σημαντικότερους στόχους μας, μια από τις σημαντικότερες δράσεις μας είναι η διασφάλιση ότι οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους ορθές πληροφορίες. Είναι σημαντικό και για την προστασία των καταναλωτών και για το δικό μου χορτοφυλάκι, αλλά και σε συνεργασία με άλλους επιτρόπους. Η αξιολόγηση λοιπόν αυτών των ισχυρισμών στον τομέα των καλλιτικών είναι ένα θέμα στο οποίο χρειάζεται να αναπτύξουμε κατευθυντήριες γραμμές πολύ συγκεκριμένες, ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Με βάση το οποίο θα κρίνεται κατά πόσον ένα χειρισμός είναι αποδεκτός ή παραπλανητικός. Κατά πόσον ένα χειρισμός θέτει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. Άρα θα εστιάσουμε σε αυτό το θέμα σύντομα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που θα καθορίσει με ποιο, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογούνται αυτοί οι ισχυρισμοί. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Τελείωσε η ώρα μας εδώ. Ευχαριστώ εκείνους που έκαναν τις ερωτήσεις και ε, τον ε, οριστέντα Επίτροπο κύριο Μίμητσα για τις απαντήσεις και παραδίδω και πάλι στον κύριο Χάρμπορ. Well, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την, τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που έθεσαν και τις οποίες φυσικά θα παρακολουθήσουμε και εμείς. Και προχωράμε στον επόμενο γύρο. Ξεκινάμε τον κύριο Ρόσφορ και μετά την κυρία Βανιού. Κύριε Ρόσφορ, έχετε τέσσερα λεπτά. Καλώ ήρθατε και καλώ ήρθαν και στην ευρωπαϊκή οικογένεια οι Κροάτες και όλοι οι κροατέ καταναλωτές. Θέλω να σας θέσω μια δύσκολη ερώτηση, την ερώτηση του προπολογισμού. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι ε, αρμοδιότητα της Επιτροπής, είναι κάτι που γίνεται μεταξύ του Κοινοβουλίου και μεταξύ του Συμβουλίου και φυσικά θα το σεβαστώ αυτό, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονό ότι έχετε ένα πολύ ευρύ χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινή ζωή και πολλά προγράμματα. Και λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς είστε αισιόδοξο ή απεσιόδοξο όσον αφορά την έκφαση των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό. Και δεύτερον, εάν τελικά γίνουν περικοπές, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας ποια θα είναι τα προγράμματα εκείνα που κατά προτεραιότητα εσείς θα διατηρήσετε, αλλά κυρίως ποια θα είναι εκείνα που τελικά θα αναγκαστείτε να περικόψετε, να μην τα υλοποιήσετε. Thank you very much for uh, a question related to the Σας ευχαριστώ πολύ που θέσατε το θέμα του προϋπολογισμού. Γνωρίζω ότι ξανά ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις και ευελπιστώ ότι σύντομα θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα προπολογισμό, να γνωρίζουμε και ποια είναι τα κοντήλια που έχουμε στη διάθεσή μας για την προστασία του καταναλωτή. Πράγματι υπάρχουν πολλά μικρά προγράμματα, περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως. Σήμερα η περικοπή είναι 4 5% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να συνεισφέρω στις διαπραγματεύσεις αυτές τους εξής. Θα επιδιώξω το ύψος των κονδυλίων για την προστασία του καταναλωτή να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά γίνεται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Σωστή οι περικοπές να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες, γιατί θεωρώ ότι το πρόγραμμά μας είναι ήδη ορθαορισμένο, είναι ήδη σαφές, είναι μικρό και διαχειρίσιμο. Και έτσι η διαχείριση του προγράμματος πρέπει να γίνεται αναλογικά προς το μέγεθος του προγράμματος, το, το ύψος του, της χρηματοδότησης που χρειάζεται. Εάν περικοπούν ακόμα περισσότερο τα κονδύλια, δεν θα, θα ήταν δυνατόν να υπάρξει υποστήριξη της προστασίας του καταναλωτή από ευρωπαϊκή πλευρά. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξο. Ε, είμαι αισιόδοξο ότι τελικά θα καταφέρουμε να έχουμε στη διάθεσή μας ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας του καταναλωτή που θα χρηματοδοτεί τις, ε, τους πίνακες επιδόσεων, τους ε, ε, μελέτες, τη λειτουργία ευρω, της Ευρωπαϊκής, ε, Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατανολητή. Αυτός νομίζω είναι ένας α, κοινός στόχος. Ωραία, αλλά δεν μου απαντήσατε. Τελικά ποια θα είναι τα προγράμματα που δεν θα μπορέσετε να χρηματοδοτήσετε. Εκεί είναι το πιο σημαντικό. Αλλά πιάνομαι από ένα σημείο που αναφέρατε ότι είπατε ότι είναι μια εξαιρετικά εγκάρσια πολιτική, πολύ οριζόντια πολιτική προστασία ε, ε, προστασίας του καταναλωτή που αφορά και άλλους επιτρόπους και η ερώτησή μου είναι έχετε την πρόθεση να συνεργαστείτε και με άλλους επιτρόπους δηλαδή να τους εξηγήσετε ποιες είναι οι προτεραιότητες της προστασίας του καταναλωτή και να καταλήξετε σε συνεργασίες έτσι ώστε πιθανώ να αξιοποιηθούν και προπολογισμοί και το, το μάλλον του προπολογισμού που έχω στη διάθεσή τους του ναι. μεγαλύτερα ποσά από ότι ο μικρό προπολογισμό τη προστασία του καταναλωτή. Μίμη, σε ευχαριστώ που αναφέρετε και πάλι ότι ο, τα κονδύλια για την προστασία του καταναλωτή αφορά στα κεντρικά στοιχεία της πολιτικής, τον πυρήνα της πολιτικής αυτής. δηλαδή τον τομέα εκείνων της πολιτικής προστασίας του καταναλωτή που αποτελεί αρμοδιότητα της, ε, του Επιτρόπου και της Γενικής Διεύθυνσης ε, ΣΑΝΚΟ. Ωστόσο, η προστασία του καταναλωτή δεν είναι θέμα καθετοποιημένο, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο ε, αυτές τις δραστηριότητες γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα προγράμματα σε χαρτοφυλάκια άλλων επιτρόπων που έχουν αντίκτυπο στα δικαιώματα των καταναλωτών. Άρα και από άλλου τομεί του προπολογισμού και από άλλε γραμμέ του προπολογισμού μπορούν να εξευρεθούν χρήματα για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην προστασία του καταναλωτή και θα συνεργαστώ με άλλου επιτρόπου για προ αυτή την κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ. Και τώρα η Μπερναντέτ Βαρνιό και μετά η Σάντρα Κανιέτ. Merci. Monsieur le commissaire désigné, bienvenue. Ευχαριστώ. Κύριε Οριστέντα, Επίτροπε, καλωσορίσατε κι εσείς και η πανέμορφη χώρα σας. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που δεν είναι αρμοδιότητα αποκλειστική δική σας, αλλά έχει όλο και περισσότερες επιπτώσεις στους καταναλωτές. Και αυτό είναι οι απομιμήσεις προϊόντων. Ε, είναι ένας ε, τομέας πολύ επικερδές, σύμφωνα με τον ΩΣΑ, αποφέρει 300 δις ευρώ το χρόνο. Βεβαίως, σε αντίθεση με τα κλασικά προϊόντα ε, που είναι απομιμήσεις ε, είναι και επικίνδυνα ε, τα φάρμακα, τα τρόφιμα, ηλεκτρικές συσκευές, καπνός, παιχνίδια, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ένα τρίτο των κατασχέσεων στα τελωνία. Μάστιγα ολόκληρη και τι συγκεκριμένες δράσεις προτίθεστε να λάβετε για την ενημέρωση κυρίως των καταναλωτών και μάλιστα των πιο ευάλωτων. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. που αναφέρεστε σε αυτό το πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο ζήτημα προστασίας των καταναλωτών. Ναι, η απομίμηση προϊόντων είναι απειλή ε, προς τους καταναλωτές. Στην καλύτερη περίπτωση επειδή είναι πλαστά, αλλά στη χειρότερη περίπτωση πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι μόνο αν είναι μαϊμού το προϊόν ή όχι, αλλά ε, αν είναι ασφαλές ή όχι ε, να κυκλοφορεί στην αγορά και μπορεί κανείς να ταυτοποιήσει πολλά προϊόντα σε πολλούς τομείς που κυκλοφορούν στην αγορά και είναι πλαστά. Κυρίως ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την τεχνική ασφάλεια του αυτοκινήτου ή και παιχνίδια επίσης. Μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο και μεγαλύτερη απειλή για την υγεία των ε, παιδιών, ακόμα και την ίδια τη ζωή ε, του καταναλωτή σε μικρή ηλικία. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους τους ενεχομένους και ε, όλους όσοι είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια των προϊόντων. Και ένας από αυτούς θα είμαι και εγώ εφόσον με επιβεβαιώσετε και διοριστώ. Βλέπω λοιπόν σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους επιτρόπους, τον κύριο Σεμετά ας πούμε, που είναι για τους τελωνιακούς ελέγχους, η Μπαρνιέ για την πνευματική ιδιοκτησία, ή με τον αντιπρόεδρο Ταγιάννη για την ε, βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, για να καταπολεμήσουμε την αυξανόμενη αυτή τάση απομιμήσεων προϊόντων. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν εμείς, να ε, προλαμβάνουν τα τελωνία τα προϊόντα αυτά να μην κυκλοφορούν στην αγορά όπως είπαμε και επίσης να βελτιώνεται η χνηλασιμότητα αυτών των προϊόντων στην αγορά για να μπορούν να ε, αποσύρονται με όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πολύ συγκεκριμένα κύριε Επίτροπε, ποιε συνέργειε θέλετε να αναπτύξετε με τους υπόλείπου επιτρόπους ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου αλλά και για συντονισμένη δράση απέναντι σε τρίτες χώρε. Yes, ναι, Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμπληρωματική ερώτηση. Και διευρύνει πραγματικά το πλαίσιο εκείνων που θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης των ε, παραποιημένων προϊόντων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπάθησα να εξηγήσω ε, ποια θα μπορούσε να είναι η κοινή δράση, αλλά Βεβαίως εξαρτάται πάρα πολύ από τις ε, εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου, είτε πρόκειται για τελωνιακές αρχές, εποπτικές της αγοράς ή αρχές ε, που ασχολούνται με την ιχνή λασιμότητα των προϊόντων. Θα ήθελα και πάλι να πω ότι το στοιχείο της συνεργασίας και προτεραιότητα για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα του αρμοδίου επιτρόπου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ε, συνεργασία με τις εθνικές αρχές για τα ε, προϊόντα αυτά της απομιμήσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καλνιέτε και μετά ο κύριος Γκαρσές Ραμών. Υποψήφιοι Επίτροπε, θέλω να σας συγχαρώ, να σας ευχηθώ και καλό κουράγιο, γιατί ξέρω πως αυτή η ακρόαση είναι βασανιστήριο για τον οριστέντα Επίτροπο κάθε φορά. Ωστόσο θα ήθελα να συνεχίσω μετά από αυτά που ρώτησε ο κύριος Βάμπα στην αρχή της σημερινής ακρόασης. Η απάντησή σας, στην απάντησή σας δεν αναφέρατε σαφή προτεραιότητες για το τι θα εφαρμόσετε στην ε, ατζέντα για τον καταναλωτή. Και πάλι λοιπόν θα επαναλάβω την ίδια ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε δύο, τρεις, τρία νομοθετικά κείμενα που θα είναι η δική σας προτεραιότητα για την επόμενη σύντομη περίοδο, τη δεκάμενη περίοδο των 12 μηνών και έπειτα γιατί οι συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στις συγκεκριμένες νομοθετικές δράσεις που μπορεί θα πρέπει να λυθούν, να αναλυθούν στη διάρκεια αυτής της σύντομης 16η περίοδου. Ε, όσον αφορά το νομοθετικό έργο που θα είναι της άμεσης αρμοδιότητά μου, τη άμεση ευθύνης μου, ε, έχω την εντύπωση πως η νομοθεσία που ήδη είναι στη διαδικασία μπορεί να αρκεί ώστε να καλύψει την ασφάλεια των προϊόντων, την εποπτεία της αγοράς και το συντονισμό αυτής, καθώς και την βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών στις κλιματοπιστωτικές υπηρεσίες τους μέσω των λογαριασμών τους. Εάν μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις νομοθετικές ε, διατάξεις, προτάσεις μάλλον, ε, μέσα στη διάρκεια αυτής της σύντομης θητείας θα συμβάλλουμε πολύ στην πολιτική για τον καταναλωτή. Γι' αυτό δεν προβλέπω αυτή τη στιγμή κάποιες ε, σπουδές νομοθετικές προτάσεις που να προκύπτουν από το πεδίο των άμεσων μελλοντικών μου ε, αρμοδιοτήτων. Όμως γι' αυτό είναι αυτή η τομές, οι τομείς των ε, δικαιωμάτων του καταναλωτή. Να δούμε δηλαδή την εφαρμογή, για παράδειγμα, τις οδηγίες ε, για την καταναλωτική πίστη, να δούμε ποια είναι η εφαρμογή των ε, αθέμητων εμπορικών πρακτικών, προστασία των δεδομένων στο ίντερνετ, αν όντω προστατεύονται καλύτερα, ε, ουδετερότητα μέσω των νομοθετικών προτάσεων που θα φτάσουν σύντομα στο Κοινοβούλιο. Εγώ βλέπω το ρόλο μου ως ε, την επιβολή του, της προοπτικής του καταναλωτή σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις για τους επόμενους μήνες που, και θα είναι αρκετή εργασία αυτή για την επόμενη περίοδο. Σας ευχαριστώ. Εγώ... Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την ουδετερότητα του διαδικτύου που μόλις αναφέρατε, αναφέρατε. Θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς τι εννοείτε. Εννοείτε την εφαρμογή του πακέτου τηλεπικοινωνιών μόνο, διότι το ΕΛΚ και το Ευρωκοινοβούλιο είναι κατά οποιασδήποτε νέας νομοθεσίας που θα επεκτείνει το θέμα αυτό σε άλλα προβλήματα για την οδετερότητα του διαδικτύου, τουλάχιστον κατά αυτή την νομοθετική περίοδο αυτή τη ε, σας ευχαριστώ πολύ για το ότι τονίσατε την ε, επιγραμμική πολιτική για τον καταναλωτή που διαρκώς ε, αυξάνεται. Είναι όντως αλήθεια ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στις επιγραμμακές συναλλαγές. Φυσικά είναι μια, ένας τομέας πολιτικής όπου είναι επικεφαλής η Αντιπρόεδρος Κρούς και στην προετοιμασία για την ακρόαση μπόρεσα να έχω μια πρώτη εικόνα των των κύριων αξώνων ε, της επερχόμενης πρότασης, αλλά από ό,τι κατάλαβα πρόκειται για μια πρόταση που θα ασχοληθεί με το θέμα της ενιαίας, αγορά αγοράς για τις τηλεπικοινωνίες και την πτυχή της ουδετερότητας ε, των επιγραμμικών αγορών για τους καταναλωτές, αλλά παρακαλώ να έχω λίγο περισσότερο χρόνο για να εξετάσω και τις λεπτομέρειες. Uh, uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Καρσές Ραμόν και μετά ο κύριος Κάρας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μιμίτσα, για την παρουσία σας σήμερα ενώπιον μας, που έρχεστε από αυτή την πανέμορφη χώρα της Κροατία. Στην αρχική σας τοποθέτηση μου άρεσαν πολύ αυτά που είπατε ε, για τους καταναλωτές ε, που τους αντιλαμβάνεστε ως πολίτες και ότι έχουν μεγάλο ειδικό βάρος στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τα πράγματα και πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση με τη βοήθειά τους, με τόνωση της εσωτερικής ζήτησης που θα έρθει από τους καταναλωτές. Θα πρέπει επίσης οι αγορές να είναι στην υπηρεσία των καταναλωτών και όχι το αντίστροφο. Αυτές λοιπόν ε, οι απόψεις σας νομίζω προσανατολίζονται προς μια καλή πολιτική κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας και των ευθυνών σας. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις πολύ σύντομα. Πρώτον, πώς αντιλαμβάνεστε την ανάπτυξη της νέας ατζέντα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή που πρόκειται να εγκριθεί προσεχώς από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης πώς βλέπετε την απαραίτητη εφαρμογή της αρχής προφύλαξης για θέματα τόσο ευαίσθητα για τους καταναλωτές όπως είναι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και τα προϊόντα νανοτεχνολογίας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γασές Ραμόν. Σχετικά με την έκθεση για την αναθεώρηση της ατζέντα ε, των καταναλωτών, πρέπει να σας πω ότι θα έρθει πολύ σύντομα στο Κοινοβούλιο και θα είναι καταπληκτική ευκαιρία για όλους μας να μπούμε σε ουσιαστική συζήτηση για ε, τα επιτεύγματα μέχρι τώρα, για τις μέχρι τώρα εξελίξεις, ε, ε, με έναν τρόπο συνολικό, για να δούμε ποιες είναι οι συνολικές προκλήσεις, όλοι οι πυλώνες αυτής της ατζέντας. Προσβέλεπω λοιπόν στη συζήτηση αυτή ε, που θα αρχίσει πολύ σύντομα με το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα και τα θετικά και τα ωφέλη από την ατζέντα αλλά και όσες δράσεις χρειάζονται και εκκρεμούν ακόμα. Πώς θα βελτιωθεί, αυτό θα πρέπει να εντοπίσουμε και ε, με ποιο τρόπο θα γίνουν όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι Ο κύριος κορμός αυτής της ατζέντα ε, ήδη έχει ολοκληρωθεί, αλλά θα πρέπει να στοιχηθεί κάπως με την πραγματικότητα και με τις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι αγορές. Και αυτό έχει να κάνει και με την ε, αυξανόμενη ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό χώρο γέννη, αλλά και με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στους καταναλωτές, όπως και γενικά την παγκοσμιοποίηση των αγορών με παγκόσμιους πρωταγωνιστές που επηρεάζουν και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά λοιπόν και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας προς την κατεύθυνση αυτή. Έχετε συμπληρωματική κύριε Γαρσές ή όχι. Ναι, ευχαριστώ. Σε σχέση μόνο με την αρχή της προφύλαξης και τα ευαίσθητα προϊόντα για τους καταναλωτές. Όπως είπα, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας. Θα ήθελα να μάθω την άποψή σας και να σας ενθαρρύνω οπωσδήποτε να δείξετε σθένος ε, στην υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ε, yes, indeed, when... Ναι. Όταν μιλούμε για αυτές τις νέες πραγματικότητες στην αγορά, γενικώ στην εσωτερική αγορά ερχόμαστε αμέσως αντιμέτωποι με την αρχή της προφύλαξης. Δηλαδή, ανάλυση κινδύνου. Καλύτερα θα πρέπει να γίνεται αυτή έτσι ώστε να έχουμε πάντα στο επίκεντρο της προσοχής την προστασία των καταναλωτών σε νέα τμήματα της αγοράς, σε νέες συνθήκες της αγοράς, ε, με την ίδια ισχύ όπως ε, υπήρχε προστασία στις κλασικές αγορές. Η ασφάλεια των προϊόντων στη σύγχρονη αγορά δεν είναι καθόλου δεδομένη. Θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε αυτή την ε, ασφάλεια με μέτρα προφύλαξης, για να δούμε ποιες είναι οι λύσεις που θα αντέχουν και στο μέλλον για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες και τις προσδοκίες αλλά και τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών. Βεβαίως, θα ε, προβούμε και σε εκτίμηση κινδύνου και σε προφυλάξεις σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και, και αυτές που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας. Ο κύριος Κάρας, τελευταίος ομιλητής σε αυτό το γύρο των ερωτήσεων. Κύριε Οριστέντα Επίτροπε, θα κατανοήσετε ότι ως Αυστριακός και Ευρωπαίος χαίρομαι που την 1η Ιουλίου ε, ε, προσχωρεί στην Ένωση η Κροατία. Αλλά ακούω αυτές τις δύο ώρες τη συζήτηση και δεν φταίτε εσείς. Ε, και όλο και περισσότερο αμφιβάλλω αν είναι σωστό ε, να αυξάνεται συνεχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ακούμε ότι είναι συναρμοδιότητες, εγκάρσιες στη διοίκηση και σας ερωτώ. Εσείς αισθάνεστε άνετα που βγαίνει έτσι ξεχωριστά η προστασία των καταναλωτών, ενώ είναι αρμόδιοι τόσο πολλοί επίτροποι και τόσες υπηρεσίες, θα κάνετε μια task force όλων των επιτρόπων που είναι αρμόδιοι για την προστασία των καταναλωτών, για να συντονίζονται και όλες οι γενικές διευθύνσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, εσείς είστε διπλωμάτης, αλλά χρειαζόμαστε και περισσότερους ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι τρεις μεγαλύτερες αδυναμίες του φακέλου σας, του χαρτοφυλακίου, της προστασίας των καταναλωτών και ε, τι πρωτοβουλίες ε, θα λάβετε πέρα των όσων ήδη είναι επιτάπητος για να ξεπεραστούν αυτές οι αδυναμίες. Thank you very much, Mr. Karas, for... Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάρας Πολύ σημαντική αυτή η πτυχή που θέσατε ως προς την αποτελεσματικότητα αλλά και το πεδίο του χαρτοφυλακίου της ε, πολιτικής καταναλωτών. Κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι πραγματικά που η πολιτική καταναλωτών είναι ένα θέμα για το οποίο έχουν αρμοδιότητα πολλοί επιτροποί. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η ισχύση, τουλάχιστον θα μπορούσε να αποτελέσει η ισχύ της πολιτικής καταναλωτών. Αν ο καθένας ε, δίδει αντίστοιχη σημασία και αφιερώνει τον ίδιο χρόνο και την ίδια ενέργεια σε αυτά τα θέματα των καταναλωτών. Αν όλοι οι επίτροποι έχουν την ίδια προσέγγιση. Εκινώντας λοιπόν από αυτή την κάθετη δομή και την άσχετη, ε, τώρα δημιουργείται μια άλλη τάση. Ε, έχουμε πολιτικές που είναι πιο κοντά στον κόσμο, πιο κοντά στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά προσβλέπω και αναμένω συνεργασία ε, ε, άλλους επιτρόπους. Συνάντησα πολλούς και συμφωνήσαμε να έχουμε τακτικές επαφές και ανταλλαγή απόψεων. για το πώς θα βελτιωθεί αυτή η συλλογική δράση και η συναρμοδιότητα για τα θέματα των καταναλωτών. Δεν υπάρχουν ασθενείς, δηλαδή τι εννοώ, δεν εξασθενίζουν οι ε, πολιτικές ε, επειδή είναι σε διάφορα χαρτοφυλάκια. Το θέμα είναι να καταβάλεις κάθε δυνατή προσπάθεια και να συνενώνεις τις δυνάμεις σου για να ε, επιτυχάνεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κύριε Ρουσταντά Επίτροπε, κατά την άποψή σας, στην πολιτική προστασία των καταναλωτών, όπου χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία των καταναλωτών, για να υπάρχουν οι τέσσερις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, και να μπορούμε πλήρως να υλοποιούμε αυτό το δυναμικό. Διότι επανειλημμένα έχουμε μία αντίφαση μεταξύ της πολιτικής προστασίας των καταναλωτών και των τεσσάρων ελευθεριών. Καμιά φορά οι διαφορές στην νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών ε, οδηγούν σε εμπλοκή την ουσιαστική υλοποίηση των τεσσάρων ελευθεριών στην εσωτερική αγορά. Απάντηση. Οι τρεις προτεραιότητες που προσπαθώ να προωθήσω και τις ανέφερα εισαγωγικά, ε, εδραίωση, συντονισμός και επικοινωνία, consolidation, coordination, communication στα αγγλικά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και τα τρία με την προστασία των καταναλωτών, αλλά μπορούν να αποδειχθούν και μεγαλύτερες αδυναμίες στην προστασία των καταναλωτών, εάν δεν ε, αξιοποιηθούν και αναπτυχθούν πλήρως. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτή τη σύντομη περίοδο των 16 μηνών που απομένει να αφιερωθώ εκεί, να βελτιώσω ακριβώς την εδραίωση, τον συντονισμό και την επικοινωνία. Αυτά τα τρία C. και γενικότερα σε όλες τις πολιτικές. Ε, αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί πέρασε και ο χρόνος μου, ε, λεπτό είχα για την απάντηση μόνο. Και ε, με χαρά να τα συζητήσουμε σε περίπτωση που ε, διοριστώ να πούμε σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και να βρούμε από κοινού ένα δρόμο για τις πιο συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται. Thank καλό. Περνάμε στον πέμπτο γύρο και θέλω να δούμε τι χρόνο έχουμε λίγο στη διαθεσή μας. Ήμασταν πολύ γενναιόδοροι μέχρι στιγμή. Έχουμε ακούσει 20 ομιλητές, έχουμε 45 λεπτά στη διαθεσή μας και έχω ακόμα άλλους 11 και θέλω να μπορέσει και ο Επίτροπος να ολοκληρώσει. 5 λεπτά μισή λεπτά θα πρέπει να περιορίσουμε ε, τις ερωταπαντήσεις και παρακαλώ να είστε δηλαδή πιο σύντομοι και να πω και στον ε, οριστέντε επίτροπο ότι θα είμαι πιο αυστηρός και θα του ανάβω το κόκκινο φως νωρίτερα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουμε. Ε, φαντάζομαι πως μπορώ να βασιστώ και στη δική σας ε, ανοχή, αλλά παρακαλώ να, πιέσετε, να θέσετε δύσκολες ερωτήσεις και να πιέσετε και για τις απαντήσεις. Έχουμε το πέμπτο γύρο που πάει Στάιλερ. Uh, Mr. De Jong for a second time, so I hope you'll be extremely brief, um, and Mr. Obermeyer. Uh, so we start with Mr. Poupakis. Ε, ξεκινάμε τον κύριο Πουπάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Σύμφωνα με το, θα ήθελα την άποψή σα. Σύμφωνα με το τελευταίο βαθμολόγιο για του καταναλωτέ, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονό των υψηλών αποκλήσεων στι τιμέ προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών, χωρί να σχετίζεται μάλιστα με την αγοραστική δύναμή του. Αυτό δείχνει ότι οι καταναλωτέ στι λιγότερε εύπορε χώρε πληρώνουν σχετικά υψηλότερε τιμέ. Χαρακτηριστικά θα ήθελα να αναφέρω ότι, παράδειγμα, στη χώρα μου την Ελλάδα, έπειτα από 6 χρόνια ύφηση και 25% μείωση του ΑΕΠ, βασικά αγαθά καθημερινή ανάγκη και διατροφή πολλούνται σε πολύ υψηλότερε τιμέ σε σύγκριση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, όπου το μέσο εισόδημα εκεί είναι υπερδιπλάσιο. Έχοντα λοιπόν σαν δεδομένο ότι η δικαιολόγητη απόκριση τιμών μπορεί να είναι ένδειξη λειτουργία και κερματισμού τη αγορά και ότι οι καταναλωτικέ οργανώσει κάνουν λόγο για παιχνίδια των πολυεθνικών στο ράφι, θα ήθελα να ρωτήσω πώ εξηγείται τέτοιου είδου αποκλήσει στι τιμέ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη, και αν θεωρείτε ότι αποτελούν ένδειξη δυσλειτουργία και κατακαιρματισμού τη αγορά και αν μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτά. Ευχαριστώ. Yes, thank you very much, Mr. for this question. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πουπάκη για αυτήν την ερώτηση που όντως ε, περνά στην καρδιά, ε, αφορά την καρδιά της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να λειτουργεί πλήρως η εσωτερική αγορά κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής και ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης και δεν είναι διόλου εύκολο να λειτουργεί όταν η κρίση είναι άνισα μοιρασμένη στην ιστορική αγορά, ώστε δηλαδή κάποια κράτη-μέλη, κάποια τμήματα μάλλον της αγοράς να, είναι πιο, να επηρεάζονται περισσότερο από τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης, ενώ άλλα λιγότερο. Γι' το λόγο έχουμε την ενιαία πράξη και γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή αλλά και τα ίδια τα κρατημέλη πρέπει να προσπαθήσουν να έρθουν όσο γίνεται πιο κοντά στη, στα θεμέλια της ευρωπαϊκής αγοράς το θέμα του ευάλωτου χαρακτήρα θα πρέπει να ερευνηθεί σύντομα από τις, επιτροπές, ε, από τις υπηρεσίες της Επιτροπής είτε πρόκειται για ευάλωτο χαρακτήρα λόγω του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης ε, είτε πρόκειται για ευάλωτο χαρακτήρα λόγω ηλικίας ή άλλους λόγους, πρόκειται για άλλους λόγους. Εν βαση περιπτώσει μια συλλογική συγκέντρωση πληροφοριών ώστε να έρθουμε πιο κοντά στην ίδια την έννοια της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, συμπληρωματικά θα ήθελα να επιμείνω. Με δεδομένο ότι οι τιμέ συγκαταλέγονται στι κύριε ανησυχίε των καταναλωτών και αποτελούν κύριο και καθοριστικό παράγοντα τη ευημερία του, πιστεύετε προσωπικά ότι η ύπαρξη ενό ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου τιμών θα μπορούσε να συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών και στον περιορισμό κερδοσκοπικών πρακτικών. Εν γέννη θα έλεγα ότι το να εμβαθύνει κανείς στο θέμα της ρύθμισης τιμών ή της παρέμβαση τιμών δεν είναι ε, έννοια που ανήκει στην εσωτερική αγορά ή στην ελεύθερη αγορά. Ωστόσο, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε και να κάνουμε μάλλον κατά την απόψή μου είναι ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διάλογο υψηλού επίπεδου ανάμεσα στους διάφορους επιτρόπους και τους διάφορους φορείς ώστε να εξετάσουμε το θέμα αυτό και να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιες πιο αναλυτικές μελέτες ε, για το θέμα, να δούμε ποιες είναι, θα είναι οι συστάσεις και το πλαίσιο ώστε το πρόβλημα αυτό να μπει στην καρδιά της πολιτικής στην Ευρώπη έτσι ώστε να αυληθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στην αγορά όσο γίνεται. κυρία Στάιλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Ε, θα ήθελα εγώ να μιλήσω για το ηλεκτρονικό βιβλίο και την πρόσβαση στις βιβλιοθήκες. Αυτή τη στιγμή πολλές βιβλιοθήκες ε, δεν μπορούν να βάλουν ε, τα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή στο δίκτυο επειδή οι εκδότες δεν δίνουν τις άδειες. Ε, εφόσον βλέπουμε λοιπόν αυτή την επανάσταση ε, δεν μπορούμε να βλέπουμε με την ψηφιακή επανάσταση να επιτρέπεται μόνο για όσους έχουν τα μέσα ε, για να την παρακολουθήσουν. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο διαχωρισμό. Τι δράση μπορείτε να κάνετε με τον επίτροπο που έχει αυτό το ρόλο, ε, ως επίτροπος μάλλον που έχετε μια οριζόντια εγκάρσια εντολή μαζί με τους 11 επιτρόπους με τους πρέπει να συνεργαστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ που αναφέρατε το θέμα των ηλεκτρονικών βιβλίων εν γέννη την ηλεκτρονική αγορά για τους καταναλωτές. Η αυξημένη χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων αντικατοπτρίζει την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία των ψηφιακών προϊόντων εν γέννη. Για τους καταναλωτές και γι' αυτό πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ψηφιακή αγορά για τους καταναλωτές. Και όταν ε, μιλάμε για το ηλεκτρονικό βιβλίο, διαπιστώνσαμε τα τελευταία χρόνια την αύξηση των τιμών των ηλεκτρών βιβλίων λόγω, θα έλεγα, της αλλαγής της πρακτικής των μεγαλύτερων εκδοτών και φορέων που μετακινήθηκαν από το είδος συμφωνίας που είχαν. Μετακινήθηκαν δηλαδή από τη μια μέθοδο ή ένα μοντέλο σε άλλο. Και αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Αντιπρόεδρος Αλμούνια στον τομέα του ανταγωνισμού είναι να πάρει τις, δεσμευτικές, τις δεσμεύσεις μάλλον των μεγάλων εκδοτών να επανέλθει στην έννοια του χοντρικού εμπορίου της συμφωνίας αυτή ώστε να μπορέσει να μειώσει τις τιμές των ηλεκτρονικών βιβλίων μέσα σε μια κάποια χρονική περίοδο και αυτό είναι και το πραγματικό συμφέρον του καταναλωτή ώστε να μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιλογή και να υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός στην αγορά. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε στην Κομισιόν. Εμείς θα μπορούσαμε και συνδεόμαστε ήδη με τις διάφορε δράσεις. Η μία είναι ε, άδεια για την Ευρώπη, License for Europe, και αφορά τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα των ηλεκτρονικών βιβλίων, αλλά μεταξύ άλλων, αλλά και ένα ουσιαστικό δίκαιο για τα για τα copyrights, φαντάζομαι πως έτσι θα καλύψουμε αυτή τη διαδικασία. Thank you, Commissioner, for that, that, answer. And I think uh, you commit... Σας ευχαριστώ για αυτή την απάντηση και για την ε, δέσμευσή σας. Είναι ένας πολύ σημαντικός δημόσιος χώρος οι βιβλιοθήκες. Έχουμε βιβλιοθήκες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτές έχουμε πρόσβαση. Αυτή η πρόσβαση στη γνώση είναι πολύ σημαντική. Και σε σχέση με το τι θα κάνετε για τους ευάλωτους καταναλωτές, ε, τι θα κάνετε μάλλον τους ευάλωτους καταναλωτές ε, μέσα στο πλαίσιο αυτής της ψηφιακής επανάστασης, ώστε να μείνουν πίσω. Επανέρχομαι για τρίτη φορά έχω την εντύπωση για τη μελέτη που θα ξεκινήσει για τη χαρτογράφηση των μορφών ε, ευαισθησίας ή ευάλωτου χαρακτήρα ομάδων καταναλωτών. Η ψηφιακή αγορά είναι ένας από τους ε, τρεις τομείς κλειδιά στην ανάλυση του αντικτύπου στις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών. Χρηματοπιστωτική αγορά, ψηφιακή αγορά. Σύντομα θα έχουμε λοιπόν πολύ καλά στοιχεία με βάση την έρευνα που θα μας επιτρέψει να προβούμε σε περαιτέρω βήματα για να αντιμετωπίσουμε τα εισεβάλλοντες ομάδες στο ψηφιακό τομέα. Κυρία Μετσόλα. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται στους καταναλωτές ε, ε, πληροφορίες ε, ώστε να διευκολύνεται η, ενημέρωσή τους. Στον τριμερή διάλογο για τα προγράμματα του καταναλωτή, το ΕΛΚΑ έχει πιέσει για τη χρηματοδότηση δράσεων όσον αφορά τα site ε, σύγκρισης τιμών. Αυτά τα site ε, αυτή η ιστοτοπή είναι πολύ χρήσιμη για να μπορέσουν οι καταναλωτές να έχουν συγκρίσιμα, αξιόπιστα, ε, εύκολα συγκρίσιμα δεδομένα. Αν και οι διαπραγματεύσει του τριμερού διαλόγου δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, χρειάζεται να αναλυφθεί δράση. Ωστόσο, η Κομισιόν έχει δείξει κάποια αντίσταση σε όλα αυτά τον τελευταίο καιρό το ερώτημα είναι, είστε δεσμευμένος να εργαστείτε με τέτοιες ε, δράσεις που θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε συγκρίσιμες ε, αξιόπιστες και προσιτές εύκολα πληροφορίες. Η Κομισιόν έχει ήδη συγκεκριμένες ιδέες για πιθανές δράσεις ε, σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Thank you very much for the uh, issue. Ευχαριστώ πολύ που θέσατε αυτό το θέμα να υπάρχουν εργαλεία για σύγκριση είναι όντως αυτό σημαντικό και χρήσιμο όπλο για τους ε, καταναλωτές για να επιλέγουν ενημέρι ε, για τα τεκτενόμενα στην αγορά. Ε, γίνεται ήδη διάλογος με πολλούς ενδιαφερομένους για αυτό το θέμα, για μελλοντικές δράσεις και μέτρα που θα πρέπει να αναλυφθούν. Ήδη από τώρα έχει συμβεί αυτό στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο ίσως μπορεί να είναι οι προσεγγίσεις και μάλιστα αντιφατικές μεταξύ τους. Θα μπορούσε κανείς να κινήσει από την εθνική πλευρά και να πει ότι συγκριτικά μέσα και εργαλεία θα πρέπει να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν σε εθνικό επίπεδο, μόνο για την εχώρια αγορά κάθε φορά, για να μπορεί κανείς να επιλέγει καλύτερα ως καταναλωτής από τα μερίδια της εθνικής αγοράς ως ένα γενικότερο σύνολο της εσωτερικής. Η άλλη όμως προσέγγιση θα ήταν ίσως πανευρωπαϊκή. συγκριτικά εργαλεία για ε, όλων των προϊόντων που κυκλοφορούν ε, στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς για να προσανατολίζεται και να επιλέγει καλύτερο ο καταναλωτής. Προσωπικά εγώ θα βελτίωνα και τα δύο. Και το εθνικό αυτό συγκριτικό εργαλείο, αλλά και το ευρωπαϊκό. Δηλαδή, όλο και περισσότερο η αγορά είναι διευρωπαϊκή και με επιγραμμική κυρίως. Ε, οι καταναλωτές ψωνίζουν από το διαδίκτυο. Άρα ε, χρειάζονται άλλα αξιόπιστα εργαλεία σύγκρισης πέρα από τα εθνικά. Ε, τώρα η πανευρωπαϊκή προσέγγιση θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δαπανηρή να γίνει τώρα. Ας έχουμε αυτή την παράλληλη προσέγγιση και βλέπουμε για να μπορούν να συγκρίνουν οι καταναλωτές. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση? Ναι, έχω. Μια σύντομη θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό που μόλις είπατε. Η πιστοποίηση σημάτων για ιστοσελίδες που συγκρίνουν τις τιμές ε, είναι εγγύηση για τη λειτουργία τους και είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυτά ε, γιατί αυτό συνιστά προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Ναι και πάλι. Η ενημέρωση των καταναλωτών και αξιοπιστία ε, των ε, ιστοσελίδων, να είναι έγκυρη δηλαδή η πληροφόρηση και αληθής, είναι βεβαίως πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο και φυσικά και θέλω να το προωθήσω. Γι' αυτό και σε αυτά τα εργαλεία σύγκριση θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια πολιτική. Αυτό γίνεται με τα λεγόμενα sweep που γίνονται μετά από συντονισμό των αρμοδίων εθνικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου ε, και θα μπορούσαν να επικεντρωθούν ακριβώς αυτό, στην αξιοπιστία της εκάστοτε ιστοσελίδας που συγκρίνει οι τιμές έτσι ώστε να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό αυτά τα στοιχεία είναι αληθή και να ανακλούν την πραγματική εικόνα της αγοράς. Συγκριστημών. Thank you. Mr. Κύριος Ντεγιόγκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μίμητσα, αυτή τη φορά θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τη δική μου έκθεση για το ε, λιανικό εμπόριο. Δύο εξελίξεις βλέπουμε. Από τη μια την ψηφιακή αγορά που ε, προωθείται πολύ και από την άλλη μεγάλα περίπλοκα στοιχεία αγοράς. Κοιτάξτε πώς έχει αυτή τη στιγμή η οικονομική κρίση. Ε, τα μικρά μαγαζιά, τα καταστήματα βάζουν ε, λουκέτο συνέχεια. Αυτό δεν το θέλουν οι καταναλωτές, αλλά δεν θέλουν να κλείνουν τα μαγαζιά, αλλά οι ίδιοι θέλουν να κάνουν αγορές από το διαδίκτυο. Πώς θα γίνει αυτό και πώς θα σώσουμε τα μικρά καταστήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεγιόγκ. αν δεν σας δώσω πλήρη και συγκεκριμένη απάντηση, αυτή τη στιγμή, στο βαθμό που θα θέλατε, θα μπορούσα, αν βρείτε άλλο, να μπω σε μια γενικότερη κατεύθυνση, ε, απαντώντας στην ερώτησή σας. Ναι, ουσιαστικά η εσωτερική αγορά και πάλι θα πρέπει να εργάζεται για τους καταναλωτές, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε, αναπτύσσοντας την πρόσβαση στην αγορά ε, της αναπτυσσόμενης ε, και μάλιστα ραγδαίας δυνατότητας ε, επιγραμμικών αγορών, αυξάνουμε τη δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών και φροντίζουμε έτσι να μειώνονται και οι τιμές. Και ταυτόχρονα αυξάνεται και η προσφορά από μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Και αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος ε, των μικρών καταστημάτων, των μικρών επιχειρήσεων να φτάνουν στους καταναλωτές και να ε, τους παρέχουν τα προϊόντα. Ε, αλλάζει η αγορά σε σχέση ας πούμε με ε, τα παλαιού τύπου μικρά μαγαζιά στους δρόμους. Θα πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ψηφιακή αγορά και έτσι ε, προστατεύονται και ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πολλούν ε, σε ηλεκτρονικά καταστήματα τα προϊόντα τους. Ντένις, yeah. θέλει συμπληρωματική ερώτηση. Σε ένα λεπτό δεν προλαβαίνω. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι για κανόνες ε, χωροταξίας, πολεοδομίας, αδειοδότησης, όταν είσαι ένα δήμο, δήμος, πώς δίνεις άδεια να ανοίξει ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο ή ένα μικρό μαγαζί. Δεν θέλω να παρατείνω τη συζήτηση, αλλά υπάρχει και ένας κοινωνικός ρόλος των μικρών καταστημάτων, τον οποίο γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεν, πλην όμως δεν λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα. Thank you very much again. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Αυτό που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να σας προσφέρω στενή συνεργασία και κοινή δράση, εν μη τι κοινή ματιά για να μελετήσουμε μαζί αυτές τις διαδικασίες που πολύ σωστά επισημαίνεται ω σημαντικό στοιχείο ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αγορά. Ας συνεργαστούμε είτε με μελέτη, να αναθέσουμε καμιά μελέτη ή να βρούμε ε, το απαραίτητο πλαίσιο ε, για προτάσεις ή για πρωτοβουλίες που ε, θα ασχολούνται επίσημα και τυπικά και με αυτό το θέμα. Και είναι και προς το συμφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών. Γιατί εγώ τα βλέπω αυτά τα δύο πάντα αλληλένδετα και άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εδώ ο κύριος Σομπερμάιερ. Γιατί δεν τον βλέπω. Όχι. Ωραία, κερδίσαμε μια χρονοφυρίδα. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο γύρο. Κύριος Χατζημαρκάκης. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει της συμφωνίας μας με τον Επιτροπό να μην υπερβούμε τις τρεις ώρες. Και θέλω να του δώσω και το χρόνο να απαντήσει. Σας παρακαλώ λοιπόν αν δεν θέλετε να πείτε κάτι, οπωσδήποτε συμπροματική ερώτηση, μην κάνετε περωτήσεις. Δεν θέλω να σας πιέσω, αλλά να δούμε πώς θα χωρέσουμε αυτό στο χρόνο. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν θα κάνω συμπληρωματική ερώτηση, οπότε μπορεί να επικεντρωθεί στην απάντηση της συγκεκριμένη. Μιλήσετε πάρα πολύ για την ενημέρωση των καταναλωτών και όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτή υπάρχει από το διαδίκτυο. Τι θα γίνει αν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φραγμός στην πρόσβαση αυτής της ενημέρωσης. Αν κάποιο είναι ένα άτομο με αναπηρία, α πούμε. Έχω την τιμή να είμαι εισηγητή για νομοθεσία που αφορά αυτό το θέμα, ε, ε, για να ε, μπορούν οι φορείς του δημοσίου από τις ιστοσελίδες τους να παρέχουν πρόσβαση σε όλους και σε άτομα με αναπηρίες. Αυτή η νομοθεσία εξαιρεί όμως τον εμπορικό τομέα, τον ιδιωτικό. Και οι άνθρωποι με αναπηρίες είναι και καταναλωτές. Βέβαια όλοι οι καταναλωτές δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στι σελίδε. γι' αυτό θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το πρώτο μεγάλο εμπόδιο στην ενημέρωση. Και ρωτώ, παρόλο που αναφερθήκατε σε αυτό, το συζήτημα των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, δεν επικεντρωθήκατε ειδικά τους καταναλωτές με αναπηρίες και πόσο σημαντικό είναι για σας προσωπικά αυτό να ε, μπορούν να έχουν και εκείνη πρόσβαση στο μεγάλο πεδίο ε, της πολιτικής για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που φύγετε αυτό το θέμα. Δηλαδή το ζήτημα των καταναλωτών που για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να έχουν ε, την ε, ίδια πρόσβαση που θα έχουν οι άλλοι καταναλωτές στις πληροφορίες για την αγορά που έχουν κάποιο είδους ε, περιορισμό. Ναι, το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, εάν επιβεβαιωθώ από το Κοινοβούλιο επικυρωθώ. Θα ήθελα η έκθεση που αφορά τους δημόσιους φορείς να επεκταθεί το ζήτημα της πρόσβασης των, δημόσιο, από τις, τις των ιστοσελίδων των δημόσιων φορέων είναι σημαντικό, η πρόσβαση είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί αυτό μονάχα. και οι καταναλωτές με αναπηρία και οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε ίδιος ε, περιορισμό στην πρόσβασή τους. Σε αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να τους λαμβάνουμε υπόψη. Άρα όσον αφορά την πρόσβαση στην ψηφιακή αγορά, άρα και οποιαδήποτε άλλη αγορά, Θέλω αυτό το θέμα να συζητηθεί, να αναλυθεί. Όχι μόνο και μόνο για να αναλυθεί, αλλά για να λάβουμε δράση μετά. Όμως πριν αναλάβουμε δράση θα πρέπει να εξετάσουμε εντελεχώς ποια είναι η ενδεδειγμένη προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέλ. Grazzi, eh, nominat, eh, ευχαριστώ, κύριε Ρεστέντα Επίτροπε. Θα ήθελα να σου ρωτήσω το Ποια είναι η άποψή σας για τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά, πολύ, ε, πολλά καταστήματα τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο προτιμησιακό σε συγκεκριμένους καταναλωτές οι οποίοι ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές και αποκλείουν εκατομμύρια άλλους καταναλωτές που ίσως βρίσκονται σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να μου πείτε πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Απάντηση. Προφανώς ε, είναι, είμαι εναντίον αυτής της πρακτικής. Οποιαδήποτε διάκριση με βάση τον τόπο διαμονήσει την εθνικότητα είναι απαράδεκτη. Δημιουργεί κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς που προφανώς είναι αντίθετο με τους στόχους που έχουμε όλοι συμφωνήσει. Άρα περιορισμοί που τίθενται στην ε, ε, διανομή ενός προϊόντος που έχει αγοραστεί ε, στο διαδίκτυο ή περιορισμοί στην πληρωμή. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και περιορισμοί που πρέπει να εξαλείψουμε από την, ε, από την ενιαία αγορά και θα κάνω ό,τι μπορώ στη συνεργασία και με τους άλλους επιτρέπους για να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές. επανέρχομαι λοιπόν, μια και έχω τη δυνατότητα κύριε Οριστέντα Επιτροπέ. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα για την να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό σε ένα συγκεκριμένο μικρό νησί, πώς οι κάτοικοι αυτού του νησιού θα έχουν τη δυνατότητα να πρόσβαση στην ενιαία αγορά, στο νησί του Κόζο. Είναι ένα ωραίο νησί απαντά. Ορίστε, οριστής Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης η οικονομική δραστηριότητα, τα πλεονεκτήματα της νέας αγοράς θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Και θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα του ε, καταναλωτή να αξιοποιήσει τον ανταγωνισμό και στις μικρές απομονωμένες νησιωτικές περιοχές της ενίας αγοράς. Πρέπει επίσης να αναπτυχθούν τα διαδικτυακά καταστήματα, γιατί αυτός είναι ένας ε, καλός τρόπος για να μειωθούν οι τιμές, για να υπάρξει ανταγωνισμός και είναι και ένας τρόπος για να εξαλείψουμε τους περιορισμούς που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κύριε Ριχριστέντα Επίτροπε, ε, θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ καλώς ορίσατε στην Κροατία ε, στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά. Οφείλω να σας πω κύριε Μίμητσα ότι αυτή τη στιγμή ε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τρέφει κάποιες αμφιβολίες ως προς τη σαφήνεια και το σθένος ορισμένων ε, απαντήσεών σας σε κάποια θέματα που μας ενδιαφέρουν πολύ. Ελπίζω στην απάντησή σας τώρα να δώσετε κάποια στοιχεία συγκεκριμένων απαντήσεων και αντικειμενικών, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Σας ερωτώ λοιπόν ως ε, μέλος της ΣΥΜΚΟ, αλλά και ως μέλος της Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων ε, των Γυναικών. Γνωρίζουμε και μάλιστα πρόσφατες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δείχνουν ότι οι γυναίκες πρωταγωνιστούν στην κατανάλωση. Κατά 70% των αγορών περίπου ε, ευθύνονται. Τι γίνεται λοιπόν για τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών των 14 θα φέρει η έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το αναφέρατε κι εσείς. Ποιες είναι λοιπόν οι γενικές γραμμές ε, αυτής της έκθεσης και προς τα πού θέλετε να κατευθυνθείτε. Ενίσχυση πραγματικά των δικτύων εθνικών οργανισμών. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ενίσχυση αυτών των εθνικών αρχών και των δικτύων. Ε, πώς θα βλέπετε εσείς θα γίνουν συγκεκριμένες, επαναλαμβάνω, προτάσεις και πώς οι διάφοροι ενεχόμενοι θα ε, συμμετάσχουν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεκδίπ. Πράγματι. Μετά την προετοιμασία που έχω κάνει για την ακροασή μου και δεδομένου ότι δεν είμαι ακόμα μέλος της Επιτροπής, ίσως αυτό να έχει ως αποτέλεσμα η σαφήνεια των απαντήσεων που σας δίνω να μην είναι η ίδια με την σαφήνεια που μπορεί να ε, αντλήσει κανείς διαβάζοντας τις προτάσεις που έχει θέσει ενώπιον του Κοινοβουλίου η ίδια Επιτροπή. Αλλά, μια και μιλούμε για την νομοθετική διαδικασία στη διάρκεια της θητείας μας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας θα επιδιώκω να εξηγώ όσο το δυνατόν καλύτερα τις θέσεις της Επιτροπής, χωρίς όμως να είμαι αδιάλακτος. Θα είμαι ανοιχτό στο διάλογο και βεβαίως εάν υπάρχουν τα κατάλληλα επιχειρήματα θα επιδιώκω να βελτιώνουμε από κοινού και στη συνεργασία μαζί σας τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Τώρα, όσον αφορά την ατζέντα για τους καταναλωτές, και για το ζήτημα των, ε, της των φύλων. Ξεκινήσαμε ήδη να μελετάμε την επίπτωση του φύλου στα δικαιώματα του καταναλωτή. Από μια πρώτη, όψεω, πρώτης όψεως δεν διαπιστώνουμε και τόσους μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Άλλοι παράγοντες, άλλες μεταβλητές κοινωνικές ή δημογραφικές έχουν μεγαλύτερη επίπτωση την ε, θέση της αγοράς όπως αυτή διατυπώνεται, αντι, αντικατοπτρίζεται στους πίνακες επιδόσεων. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το ζήτημα του φύλου και στο πλαίσιο των μελετών που θα γίνουν σύντομα για τον εντοπισμό των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών και έτσι θα έχουμε περισσότερα και πιο συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μας για να δούμε με ποιον τρόπο το φύλλο ε, επηρεάζει τη θέση του καταναλωτή ή της καταναλώτριας. Μιας και δεν έχουμε και πολύ χρόνο στην διάθεσή μας, μήπως μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς να επανέλθετε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κυρία Σένα και μετά άλλοι δύο μεταξύ αυτών κυρία Ράπτη, γιατί έχουμε ξεφύγει τελείως από χρόνο. Κύριε Οριστέντα Επίτροπε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εσά και το λαό της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά κλονίζεται από ε, ειδήσει για διαφορετική ποιότητα προϊόντων, διαφόρων τύπων σημάτων από διάφορες μάρκες που κυκλοφορούν στην αγορά οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν έχουν πρόσβαση στα ίδια ποιοτικά προϊόντα ε, και πρότυπα παντού στην Ένωση. Αυτό εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές και μεταξύ άλλων σε μια έκθεση που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει αυτό το θέμα και μάλιστα αυτό συνιστά διάκριση. Ερωτώ απλούστατα, εσείς θα κάνετε τίποτα για να ε, διεξάγει έρευνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαφορετικές ποιοτικές προδιαγραφές και πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι βήματα συγκεκριμένα θα κάνετε ως Επίτροπος από μια χώρα όπου πραγματικά έχει επιβεβαιωθεί αυτό και από τα δικαστήρια ότι είναι διαφορετική η ποιότητα των προϊόντων. Σας ευχαριστώ που καλωσορίζετε την Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστώ πολύ που αναφέρετε αυτό το θέμα της ποιότητας των προϊόντων και το τονίζετε. Ναι, βεβαίως το πρώτο θέμα για μας είναι η ασφάλεια. Πρέπει να διατηρήσουμε την ασφάλεια στο επίπεδο που βρίσκεται τώρα και να το βελτιώσουμε αν γίνεται. Και έπειτα πρέπει να έχουμε και υποπαρακολούθηση τον αντίκτυπο και την, ε, των, των δράσεών μας στην ποιότητα. Δεν θα πρέπει να, να μπορούν να παραπλανηθούν οι Καταναλωτέ στην επιλογή του όσον αφορά την ποιότητα. Η ποιότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προτιμήσει του καταναλωτή στι διάφορε αγορέ, αλλά θα πρέπει πάντοτε να, σαφώς να υποδεικνύεται ε, στους καταναλωτές. Ε, θα πρότεινα να εξετάσουμε βαθύτερα αυτό το θέμα μέσω του επόμενου βαθμολογίου, ώστε να δούμε τις απόψεις και τις απαντήσεις των καταναλωτών για το ποιο επίπεδο εγγύησης και ποιότητας αναμένουν ώστε να δούμε και τι θα βάλουμε στο επόμενο βαθμολόγιο για τις δράσεις και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σάγγελο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια, ε, οριστέντα επίτροπε, ο προ το φως σας είχε αυτό το θέμα της ασφάλειας των υπηρεσιών. Και από το 2003 πολλά πράγματα δεν έγιναν, αντίθετα με άλλο τομεί όπου έγιναν ένα σωρό πράγματα. Ξέρω πως δεν είναι βέβαια δικό σας λάθος, πάντως δεν έχει σημειωθεί πρόοδο σε αυτό το τομέα. Τώρα, συγκεκριμένο τομέας είναι ε, η πυρασφάλεια στα ξενοδοχεία και αλλού, όπου ένα σωρό πεθαίνει κάθε χρόνο. Δεν λέω ότι αυτό οφείλεται στην Κομισιόν, αλλά δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο ώστε να στηρίξουμε τα θέματα πυρασφάλειας. Ώστε οι καταναλωτές να μην χάνουν τη ζωή τους. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι στο συγκεκριμένο τομέα. Και μήπως μπορείτε να μας πείτε και αν σκοπεύει να ακολουθήσει αυτή την ανακοίνωση του board, ότι δηλαδή η υγεία και η ασφάλεια θα είναι θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Το θέμα της ασφάλειας των προϊόντων είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο από ότι ο τομέας της ασφάλειας των υπηρεσιών όλοι οι επίτροποι πρέπει να ενώσουμε τις προσπαθίες μας για να κάνουμε περισσότερα σε αυτό το τομέα. Ίσως να μην είναι δικό μου λάθος για το τι έχει γίνει προηγούμενα, αλλά σίγουρα θα είναι δικό μου λάθος αν δεν γίνει τίποτα στο μέλλον. Ακόμα και αν δεν γίνει τίποτα κατά τη διάρκεια των επόμενων 16 μηνών μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Επιτροπής. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς που ήδη είναι ε, ρυθμισμένοι, ιδιαίτερα στην ε, κατάλυση που Υπάρχει χώρος για βελτίωση των νομοθετικών ε, ρυθμίσεων που αφορούν την ασφάλεια. Επίσης μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για την υπηρεσφάλεια όχι μόνο για τις υπηρεσίες αλλά και για τα προϊόντα. Δηλαδή να βελτιώσουν τα περίμαχα υλικά Ίσως να υπάρχει και κάποιος, κάποιες άλλες ουσίες που ε, επιβραδυντές της φωτιάς, εν πάση περιπτώσει εξελίξεις σε νέους τομείς γνώσης που να μπορέσουν να, ε, να βοηθήσουν σε αυτές τις δράσεις ε, της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Και μία ερώτηση μόνο τελευταία από την κυρία Ράπτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία. Κάτι πάρα πολύ απλό. Οι καταναλωτές εξαρτώνται από τις αποφάσεις πολλών επιτρόπων. Ένας από αυτούς θα είστε κι εσείς. Η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Είστε έτοιμος να συγκρουστείτε με τους συναδέλφους σας επιτρόπους για να υπερασπιστείτε περισσότερο τους καταναλωτές σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως το collective redress. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα είναι το καθήκον μου και ο τρόπος με τον οποίο θα ασκώ τα καθήκοντά μου. Θα είμαι πραγματικά ε, σκληρός και αποφασιστικός στις ε, προσδοκίες των καταναλωτών για θέματα καταναλωτών και για όλους τους άλλους ε, τομείς που έχουν να κάνουν με το συμφέρον των καταναλωτών. Οι πρώτες μου επαφές λοιπόν και συζητήσεις με πολλούς επιτρόπους και αντιπροέδρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάνουν ε, αισιόδοξο ως προς αυτό. Υπάρχει προθυμία από πλευράς όλων να μην ε, θεωρείτε το συμφέρον των καταναλωτών ότι έρχεται σε σύγκρουση με κάποιες πολιτικές διάφορους τομείς, αλλά ήδη τα μελήματα και οι προσδοκίες των καταναλωτών να ενσωματώνονται στις πολιτικές και από ό,τι φαίνεται στο παρόν στάδιο δεν είναι μια διαδικασία αυτή που ε, θα είναι, επαναλαμβάνω, σύγκρουσιακή σε σχέση με τις άλλες πολιτικές, αλλά μάλλον ε, σε συνεργασία ε, σώματων των Επιτρόπων για θέματα αυτά πολιτικής καταναλωτών. Όποτε ε, χρειαστεί μεγαλύτερη όθηση, να είστε βέβαιοι ότι θα πιέζω εγώ τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι ε, που τηρήσατε και το χρόνο σας και τις πολλές ερωτήσεις. 29 μέλη ρώτησαν που ήταν και σκληρές ερωτήσεις. Ε, σας ευχαριστώ πολύ θα παρακαλούσα τώρα τον Οριστέντα Επίτροπο να ε, δευτερολογήσει, να κάνει μια σύντομη τοποθέτηση, πεντάλεπτη για να κλείσουμε και θα του δώσω το λόγο όσο θέλει, μέχρι πέντε λεπτά όμως ε, πριν ε, λήξει αυτή η ακρόαση. Παρακαλώ, έχετε και πάλι το λόγο. Intensive, valuable σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την έντονη, ενδιαφέρουσα και ε, εξαιρετικά πολύτιμη ανταλλαγή απόψεων. Αυτή η ευκαιρία που είχαν με σήμερα να συζητήσουμε μου επιβεβαίωσε την δέσμευση που έχετε αναλάβει και τον ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή στην ενιαία αγορά, στην εσωτερική αγορά, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο καταναλωτής θα είναι εκείνος που θα φέρει την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος του καταναλωτή και η οικονομική του δύναμη είναι σημαντική. Ευελπιστώ να είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας, στο επίπεδο που αναμένεται ε, να έχει η πολιτική προστασία του καταναλωτή. Θα προσπαθήσω τώρα να σχεγραφήσω ορισμένες από τις προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου όσο πιο γρήγορα μπορώ. Χρειάζεται να θέσω προτεραιότητες. Εάν επιβεβαιωθώ, θα εργαστώ σκληρά, θα αξιοποιήσω όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα η πολιτική προστασία του καταναλωτή σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βελτιώσω στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτή την πολιτική. Θεωρώ τον εαυτό μου ε, προστάτη, το θεματοφύλακα των δικαιωμάτων του καταναλωτή και για να επιτύχω σε αυτό το έργο θα χρειαστεί συνεργασία με πολλούς με όλους όσοι επιθυμούν να κάνουν το ίδιο. Οι προτεραιότητές μου λοιπόν είναι η συνεκτικότητα, η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια, για την ασφάλεια των διαγνωστικών προϊόντων, των προϊόντων ε, διάγνωσης in vitro, καθώς επίσης και στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των τραπεζικών υπηρεσιών όπου πρέπει να προασπίσουμε τα δικαιώματα του καταναλωτή, καθώς επίσης και η ενίσχυση της νομοθεσίας και της πρακτικής για την ε, επιβολή των κανόνων από τις εθνικές αρχές και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ευελπιστώ να ήμουν σαφής και να έδειξα ε, ε, πόσο πολύ επιθυμώ την συνεργασία και πόσο πολύ επιθυμώ τη συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους προς όφελος των καταναλωτών. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες που να αντικατοπτρίζουν, που να ανταποκρίνονται μάλλον στις ανάγκες τους. αλλά και ο τομέας των επιχειρήσεων θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί, να γνωρίσει καλύτερα τον ζήτημα της προστασίας του καταναλώτη, έτσι ώστε τα δικαιώματα του καταναλωτή να προασπίζονται ήδη από την αρχή του κύκλου παραγωγής. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή έχει ε, ήδη παράγει σημαντικό έργο και προσβλέπω σε μια στενή συνεργασία μαζί σας εάν επιβεβαιωθώ. Εάν μου δώσετε την ευκαιρία να συνεργαστούμε, θα το πράξω ιδιαίτερα σε σχέση με την νομοθεσία που εκκρεμεί ενώπιον του Κοινοβουλίου και θα επιδιώξω αυτή, αυτό, το νομοθετικό έργο να ολοκληρωθεί την τη λήξη της θητείας του Κοινοβουλίου. Αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου και με μια πιο προσωπική παρατήρηση. Διαπίστωσα προσωπικά τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή στην Κροατία. Η Κροατία είναι ένα κράτος που έχει σχετικά χαμηλή συνείδωση καταναλωτική. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια να καταπτύσσουμε το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή εγώ είμαι υπέρ της εναρμόνισης αυτής της εθνικής νομοθεσίας στην Κροατία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τώρα που η Κροατία θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπω το όνειρο ε, μιας Κροατίας που θα είναι πλήρες μέλος της ενίας αγοράς να πραγματοποιείται. Εάν επιβεβαιωθώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα επιδιώξω σαφή συγκεκριμένα πραγματικά αποτελέσματα, ακριβώς δηλαδή αυτό που χρειάζονται οι καταναλωτές για να προστατεύονται τα συμφέροντά τους, τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτόν τον επικοδομητικό διάλογο. Σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας πολλές πτυχές ε, και συγκεκριμένες ε, λεπτομέρειες των μελλοντικών πολιτικών που διαμορφώνονται και που θα πρέπει να ενισχυθούν. Μα ευελπιστώ να συμμετάσχω σε αυτή τη διαδικασία μαζί με όλες τις υπηρεσίες. Well, thank you. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κύριε Οριστέντα Επίτροπε για τη συμμετοχή σας στην ακρόαση αυτή. 30 μέλη έκαναν ερωτήσει. λάθος έπεσε στον υπολογισμό μου. Ε, περίπου τηρήσαμε και το χρόνο μας, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρίσω επίσημα το πέρας της ακρόασης, αλλά πρέπει να πω ότι οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα συνεδριάσουν στις 3 η ώρα στην αίθουσα PHS 6504 ε, 054, συγγνώμη, ε, για ε, να αποφανθούμε και να συστήσουμε την πρότασή μας στη διάσκεψη των Προέδρων και στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ραντεβού για την επόμενη συνεδρίαση και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μίμητσα για την ε, ενεργητική και δραστήρια συμμετοχή του στην ακρόαση. Ευχαριστώ.